Buon pomeriggio, credo che Καλό σας απόγευμα. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε, αν και δεν είμαστε και πολλοί. Θα έχουμε ένα πολύ μακρύ απόγευμα και αποδοτικό. Ο Ρομπέρτο Βιόλα είναι ε, μαζί μας για το θέμα υπαριθμών 10 και ο κύριος Γουίλαν. Χαίρομαστε λοιπόν γιατί σήμερα μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή την πλατφόρμα Wi-Fi for You και είχαμε συνεργαστεί και με τους ε, συναδέλφους που ήταν υπεύθυνοι επί του θέματος και λέω εκπήρας ότι οι τοπικές κοινότητες και αρχές είχαν ζητήσει τη συνδρομή μας για την ανάπτυξη αυτού του προγράμματος. Χτες λοιπόν υπήρχε μεγάλη συμμετοχή για την χρήση αυτής της πλατφόρμας. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που έχουμε αυτό το πρόγραμμα στη διάθεσή μας και θα θέλαμε και εμείς να συμμετάσχουμε σε αυτή την εκκίνηση. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ρομπέρτο Βιόλα, ο οποίος έχει στη διάθεσή του 10 λεπτά περίπου για να μας μιλήσει για την εφαρμογή του Wi-Fi for You. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα και για τους συναδέλφους μου που βρισκόμαστε εδώ για να σας μιλήσουμε για αυτή την πραγματικότητα. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για την εκκίνηση αυτού του προγράμματος και τώρα έχουμε φτάσει στην υλοποίηση. Θέλω να σας πω αυτής εξ αρχής κάτι το οποίο μας εντυπωσίασε. Ξεκινήσαμε χτες με την πλατφόρμα, την πλατφόρμα αυτή. 1100 δήμοι έχουν Καταγραφή. Και σήμερα, ρώτησα τα στοιχεία ακριβώς πριν έρθω εδώ, έχουμε 4.200 δήμους. Αν λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε 88.000 ε, δήμους συνολικά, καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι 5% όλων των δήμων στην Ευρώπη έχουν ήδη καταγραφεί στην πλατφόρμα αυτή μέσα στην πρώτη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι και η απάντηση σε αυτούς, όχι βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο είχε ταχθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μα στήριξε από την πρώτη μέρα, αλλά υπήρξαν φωνές που έλεγαν ότι δεν χρειάζεται αυτή η πλατφόρμα, δεν θα είναι επιτυχής, ο κόσμος δεν θα διαφερθεί. Ε, λοιπόν, 4.200 δήμοι σε 24 ώρες. 150 πάροχοι. Το πρώτο λοιπόν που έχω να πω είναι ευχαριστώ. Ευχαριστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ευχαριστώ στην Επιτροπή σας Σίτρε, στον εισηγητή για ό,τι κάνατε. Πράγματι μας πήρε χρόνο, είναι αλήθεια, να φτιάξουμε τη δικτυακή αυτή πύλη. Ήταν η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν οργανώσαμε κάτι για να μοιράσουμε όπως τώρα vouchers στις τοπικές κοινότητες και στους ε, δήμους και να πρέπει να υπάρξει προσαρμογή των δικτύων κτλ. Αρχίσαμε τον Νοέμβριο μόνο, βέβαια, όταν ε, δημοσιοποιήθηκε και στην επίσημη εφημερίδα η τροπολογία για την ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Και έκτοτε δουλεύουμε καθημερινά με τους συναδέλφους και από τον προπολογισμό και από αλλού για να υλοποιηθεί αυτή η πλατφόρμα. Τώρα λοιπόν είμαστε πια έτοιμοι. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι το σύστημα θα αυξηθεί. Έτσι θα υπάρξουν όλο και περισσότερες υπηρεσίες που θα προσφέρονται και περισσότερες λειτουργικότητες. Και όταν θα έχει σπάσει αυτή, αυτό το φράγμα, δηλαδή θα μπορέσουμε να φτάσουμε στις τοπικές κοινότητες με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα μπορούμε Ήδη μπορούμε να το κάνουμε με τα 120 εκατομμύρια ευρώ που είναι διαθέσιμα για το Wi-Fi for you, EU, αλλά σκεφτόμαστε το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο προκειμένου να επεκταθούμε ακόμα περισσότερο και η εμπειρία αυτή να επεκταθεί. Ανάλογα βέβαια με αυτά που θα μας πείτε και εσείς από τις εμπειρίες σας και θα μας πούνε και διάφορες τοπικές κοινότητες. Κυρία Πρόεδρε, υπάρχει μια διαφάνεια που θα μπορούσαμε να σας δείξουμε, ένα βίντεο. Ε, Συνεπώς, μερικές φορές ε, τα βίντεο δείχνουν καλύτερα τα πράγματα από τα λόγια. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι κοιτώντας τι έχει γίνει αυτές τις μέρες, ότι αυτό το δίκτυο Wi-Fi σέβεται τους πολίτες. Δεν ε, πληρώνουμε τα δεδομένα τους οι πολίτες, είναι δωρεάν και τα δεδομένα προστατεύονται. Είναι οι δημόσιες αρχές που προσφέρουν το δίκτυο. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Όσον αφορά τώρα το feedback, οι οργανώσεις, το κοινό κτλ. Ε, περιμένουμε τις αντιδράσεις τους, προς το παρόν είναι ενθουσιώδης και θα θέλουμε να συνδυαστούμε και με εθνικές πρωτοβουλίες ε, για δικτυακή πύλη με τις πορτογαλικές, τις ιταλικές αρχές, με κάποιες στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές. Έχουμε επαφές που θέλουν να αρχίσουν διαρθρωμένο διάλογο. Με 120 εκατομμύρια πιστεύουμε ότι ήδη μπορούμε να κάνουμε πολλά με σεβασμό απέναντι στα δεδομένα των πολιτών. Τώρα δεν ξέρω κύριε Πρόεδρε αν θέλετε να σας πω δύο λόγια ή ο συναδελφός μου καλύτερα για την ε, εφαρμογή, την υλοποίηση και μετά Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Κύριος Βίλαν, ο οποίος είναι υπεύθυνος ε, για... και διευθυντής του δικτύου ΚΝΕΚΤ, δικτύων περιεχομένου και τεχνολογιών. Έχουμε επικεντρωθεί σε αυτό το σημείο όσο αφορά την εφαρμογή τους τελευταίους ε, μήνες και είναι κάτι το οποίο ε, κάνει αυτή την εμπειρία πολύ απλή και χωρίς προσκόμματα, όπως είδατε και στις εικόνες. Η χτεσινή σειρά, η χτεσινή εκκίνηση με προεγγραφή, με μία απλή εφαρμογή, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή στις 15 Μαΐου, αφορά ένα διανοητικό εγχείρημα το οποίο έχει τεθεί εν πολύ σε εφαρμογή. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ορισμένα μικροπροβλήματα, αλλά το σύστημα είναι λειτουργικό. Και θέλουμε να διασφαλίσουμε κάτι το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Ε, υπάρχει το σύστημα ότι όποιος προσέρχεται πρώτος έχει και πρόσβαση πρώτος, αλλά υπάρχει και γεωγραφική κατανομή στην ε, ε, επίδοση των βάουτσερ, έτσι ώστε να ε, έχουμε έναν ελάχιστο αριθμό βάουτσερ ανά κράτος μέλος, 15 δηλαδή, και ένα μέγιστο Δηλαδή κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να λάβει περισσότερο από το 8% των κουπονιών, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη και να φτάσουμε στο ε, ποθητό αποτέλεσμα το οποίο έδειξε και το βίντεο που είδατε. Ε, θα έχουμε ένα δίκτυο Wi-Fi για την Ευρώπη τη στιγμή που θα υπάρχει περιαγωγή, πλήρης περιαγωγή, όπως είπε και ο Ρομπέρτο Βιόλα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι λίγο πιο περίπλοκο μέσα στα πλαίσια των ε, τεχνολογιών επικοινωνίας και είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα τεθεί σε εφαρμογή κατά το επόμενο έτος ακριβώς όταν ο πρώτος γύρος ε, κουπονιών θα οδηγήσει σε πραγματικές εγκαταστάσεις και θα έχουμε και την πείρα των χρηστών. Έχουμε έναν προϋπολογισμό που θα επιτρέψει τη συμμετοχή 6.000 με 8.000 κοινότητες σε 24 ώρες ε, το ίμιση αυτού του προϋπολογισμού θα μπορούσε να πληρωθεί, να έχει ήδη καταναλωθεί με βάση τον ε, γεωγραφικό επιμερισμό που σας είπα και πιστεύουμε ότι ακριβώς αυτό είχε ε, προωθήσει και το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την επιτυχία της πρωτοβουλίας και ελπίζουμε να έχει και ευρύτερες επιρροές. Ο κύριος ε, Ζωρίνιο έχει το λόγο, ο οποίος ήταν και ο κύριος εισηγητής και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ και καλό σας απόγευμα. Αυτή η μέρα, η χτεσινή δηλαδή, ήταν μια ιδιαίτερα ευχάριστη ημέρα για τον εισηγητή αυτής της μεγάλης πρωτοβουλίας και θα ήθελα να σας πω όμως ότι έχω ε, μεικτά συναισθήματα και θα σας πω γιατί. Όλοι αναγνωρίζουμε τη συμβολική και πολιτική σημασία αυτής της πρωτοβουλίας. Εάν υπήρχαν ε, επιφυλάξεις, ε, όπως είπε και ο Γενικός Διευθυντής, η εγγραφή 4.200 ε, ατόμων την πρώτη μέρα στην ουσία έχει απαλείψει τις ε, επιφυλάξεις με ταχύτητα 5G και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συνεργάτες για αυτή την εργασία έτσι ώστε τάχιστα να έχουμε μία πρόταση. Ο τριμερής διάλογος ήταν επιτυχής με τη συμμετοχή του Συμβουλίου και της Επιτροπής και με τον Γέρση Μπούζεκ, τον πρόεδρό μας, έτσι ώστε να έχουμε επιτυχής πρωτοβουλίες γιατί πολλοί έλεγαν ότι τα ζητήματα που είχαμε θα ήταν αδύνατον να επιληθούν. Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες από τις χώρες και τις τοπικές κοινότητες. Γιατί τους είχαμε υποσχεθεί μία ε, διευκόλυνση της πρόσβασης με έναν απλό τρόπο, με κουπόνια, πολύ απλά δεν ξέρω γιατί χρειάζονται 18 μήνες ε, γιατί χρειάζεται τόσος καιρός ε, για μία εγκατάσταση που στοιχίζει 15.000 ευρώ. Αυτή η τεχνολογία θα μπορούσε να αλλάξει άρδιν μέσα στα επόμενους, επόμενους 18 μήνες. Γιατί 15 και όχι 20.000. Άρα θα μπορούσαν να εγγραφούν αυτές οι οντότητες ή κοινότητες με βάση το ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης. Εξαιρετικό το βίντεο που είδαμε, αλλά υπάρχει μόνο η πύλη εγγραφής, τίποτα άλλο. Είμαστε σε μηδενική βάση ως προς τα υπόλοιπα. Δηλαδή, πέρα από την πύλη δεν έχει αναπτυχθεί τίποτα άλλο. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τις εξελίξεις. Χαίρομαι γιατί ενεγράφησαν 4.200 κοινότητες και χαίρομαι που θα τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα στις 15 Μαΐου. Αλλά εδώ δεν μιλάμε μόνο για προσβάσεις, μιλάμε για χρηματοδότηση προσβάσεων με, με ένα ενιαίο μέσω μάλλον μίας ενιαίας πύλης ταυτοποίησης σε μία ενιαία πλατφόρμα. Η ανακοίνωση είναι πολύ σαφής, όπως την είδαμε και στο βίντεο, αλλά τώρα θα πρέπει να προβούμε στην πραγματική εγκατάσταση. Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση. Πιστεύω ότι με το επόμενο πρόγραμμα στήριξης θα έχουμε μεγαλύτερη χρηματοδότηση και μπορώ να πω ότι στη χώρα μου με την βοήθεια των διαρθρωτικών ε, ταμείων μπορέσαμε να αναπτύξουμε αυτό το πλαίσιο. Θέλουν πάρα πολλές κοινότητες να συμμετάσχουν και γι' αυτό θα πρέπει να επιταχύνουμε την εφαρμογή του 5G και να μην χρησιμοποιήσουμε την ταχύτητα που είχαμε μέχρι τώρα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν θα ένιωθα καλά αν δεν σας έλεγα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και πάλι συγχαρητήρια όμως. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Ζωρίνιο και για την ειλικρίνειά του κυρίως. Ε, οι ομάδες έχουν τώρα το λόγο. Ο κύριος Μπόνι. Καταρχά ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρωτοβουλία που έλαβε εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα. Πολύ καλή. Ευχαριστούμε τον Κάρλος Ζουρίνιο, τον εισηγητή μας, διότι συζητήσαμε λύσεις, συζητήσαμε απλές λύσεις για να είναι πολύ πιο προσβάσιμο όλα αυτά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ για αυτήν την καταπληκτική έναρξη. Καταπληκτικός αριθμός δήμων και κοινοτήτων που ε, έδειξε ενδιαφέρον για να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε επίσης και για όλη αυτή την ενημέρωση που έχουμε λάβει για αυτό το πρόγραμμα και για το σύντομο βίντεο άριστη παρουσίασή του. Έχω όμως δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πώς θα αξιολογήσουμε την εφαρμογή του προγράμματος σε κάποια κατάλληλη στιγμή, γιατί θα πρέπει να μάθουμε πολύ περισσότερο για το πώς θα λειτουργήσει και για τις τεχνικές παραμέτρους και πώς θα μπορούσε να αλλάξει τη στάση των συμπολιτών μας και την διάθεσή τους να χρησιμοποιούν σε δημόσιους χώρους το ίντερνετ στο Δήμο τους ή σε οποιοδήποτε Δήμο. Δεύτερον, τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Έχουμε 120 εκατομμύρια για αυτό το εγχείρημα. Αλλά τώρα συζητάμε ψηφιακά θέματα για τους μελλοντικού ενωσιακούς προϋπολογισμούς. Πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση. Πρέπει δηλαδή να κινητοποιηθούμε όλοι. Παρακαλούμε τις ε, κοινότητες να δώσουν μια νέα υπηρεσία προς τους ε, πολίτες. Και όπως είπε και ο Κάρλος, στο μέλλον θα συζητήσουμε και ειδικές τεχνικές παραμέτρους ε, ούτως ώστε να έχουμε Wi-Fi 5G στους δημόσιους χώρους. Με βάση την πείρα σας, ε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε συγκεκριμένα να κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, και στα πλαίσια ακριβώς της συζήτησης για τη μελλοντική πρικοδότηση τέτοιων εγχειρημάτων. Ευχαριστώ. Ε, Τερέζα Γκρίφιν. Ευχαριστώ, Πατσίσιο. Αυτό είναι θέμα ισότητας. Και αν δείτε πώς αντέδρασαν οι πολίτες μας από τότε για παράδειγμα που καταργήσαμε τη, τα τέλη περιαγωγής. Είναι κάτι που επηρεάζει την καθημερινότητα των ε, συμπολιτών μας. Αυτές οι 4.000 τόσες ε, προεγραφές είναι θαυμάσιο επίτευγμα. Πολύ χάρηκα στο βίντεο, είχατε και γυναίκες δημάρχους, όχι μόνο άντρες. Και ότι συνδέσατε το θέμα με την ηλεκτρονική υγεία, e-health. Γιατί όλο και περισσότερο έχουμε ηλιοκεμένα άτομα ή άτομα με χρόνιες ασθένειες που ε, μπορούν να βοηθηθούν ή που θα χρειαστεί να βοηθηθούν με ψηφιακές μεθόδους πρόσβασης σε κάποιες υπηρεσίες υγείας που δεν μπορούν τώρα. Πρέπει να σταματήσει λοιπόν ε, να σταματήσουν αυτές οι ψηφιακές διακρίσεις. Λοιπόν, τόσο αυτό το σύστημα, όποιος πρώτος δηλώσει, πρώτος θα εξυπηρετηθεί. Θα καταφέρουμε να φτάσουμε και σε δήμους ε, που είναι πιο φτωχοί, πιο απομονωμένες κοινότητες υπαίθρου, για παράδειγμα. Έχουμε ένα μηχανισμό για να μπορέσουμε μετά να αξιολογήσουμε ποιοι συμμετέχουν. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, υπάρχει και ένα θέμα πόρων. Αν έχουμε ήδη μοιράσει τα μισά κουπόνια, η βάουτσερ, τι πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε να υπάρξουν και περαιτέρω πόροι. Και να επανέλθω σε αυτό που είπε ο Κάρλος και τον ε, συγχαίρω ιδιαίτερα για τη θαυμάσια εργασία που έκανε. Την εκτιμώ ιδιαίτερα και τη δουλειά που έκανε στην Πορτογαλία για ψηφιακά θέματα, για πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες. Το ίντερνετ πρέπει να είναι για τους πολίτες, για όλους τους ανθρώπους, όχι το ίντερνετ των πραγμάτων. Αυτό είναι ζωτική σημασία σε αυτό που κάνουμε. Και όπως και ο Κάρλος, ανησυχώ ε, για το πώς θα αξιολογήσουμε την εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Τέρεζα για τις παρατηρήσεις σου. Τελίτσκα, από το Άλντε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ευχαριστώ και τις ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις. Ως και όδης, χαίρομαι ιδιαίτερα που επιτέλους ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα. Συμφωνώ και με τον συνάδελφο Ζουρίνιο ότι μας πήρε περισσότερο χρόνο η έναρξή του. Και δεν λέω ότι φταίει μόνο η Επιτροπή, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Πάνω από 4.000 δήμοι. Πολύ καλό. Άρα ήταν απόλυτα χρήσιμη η πρωτοβουλία. Και διαψεύδονται και αυτοί που λέγανε μπα δεν θα τον παρήδησε κανείς. Αλλά έχουμε συγκεκριμένο αριθμό κουπονιών. Άρα θα απογοητεύσουμε χιλιάδες δήμους. Άρα πρέπει να κάνουμε και μια δουλειά ενημέρωσης από την Κομισιόν και από μας, γιατί κάποιοι δήμοι και κοινότητες που θεωρούν ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν, δεν θα συμπεριληφθούν. Γι' αυτό ας μην ε, καταλήξουμε ήδη, ας μην προκαταλάβουμε το πόσο έχει ήδη επιτύχει αυτό το πρόγραμμα. Τώρα εστιάζουμε στον αριθμό αιτήσεων που έχουμε και στα κονδύλια που έχουμε. Τώρα το θέμα είναι τι επίδραση θα έχει, πώς θα αλλάξει την κατάσταση. Σας παρακαλώ να επανέλθετε στην Επιτροπή μας με την αξιολόγηση τη εφαρμογή. Και θυμηθείτε πώς ξεκίνησε η συζήτηση για το θέμα αυτό. Ορισμένες πολιτικές ομάδες και ορισμένοι βουλευτές ήταν απρόθυμοι. Και πολλοί, συμπεριλαμβανομένου και του υποφαινομένου, είπα, είπαμε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Θα ήταν ένα κίνητρο για να γίνουν αλλαγές στην οτροπία, στη, στον πολιτικό πολιτισμό και στην διάθεση, την όρεξη για να αλλάξει το ψηφιακό τοπίο. Δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο κρατών μελών. Όχι, πρέπει να γίνει σε ενωσιακό επίπεδο. Αυτό πρέπει να αναλύσουμε. Τι κίνητρο δώσαμε. Εδώ θα φανεί και ρόλο τη Επιτροπή. Όχι μόνο να προτείνει συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά αυτό να οδηγήσει σε μια ολόκληρη χιονοστιβάδα αλλαγών, να αλλάξει εντελώ το περιβάλλον. Αν είμαι για παράδειγμα κάπου δήμο, εγώ δήμαρχο κάπου που δεν έγινε δεν, που δεν έκανε έτσι να συμμετάσχει. Και άμα βλέπω ότι στο διπλανό Δήμο εφαρμόστηκε και ε, είχε μεγάλες, ε, επέφερε μεγάλες αλλαγές στο διπλανό Δήμο, τότε θα θελήσω κι εγώ ακόμη και αν δεν έχω ε, αυτή την ενωσιακή χρηματοδότηση να εισαγάγω κάτι τέτοιο από το δικό μου προπολογισμό, του χωριού μου. Αυτό μπορεί να γίνει λοιπόν. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό. Οπότε, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, Ίσως θα έπρεπε ήδη να προτείνετε την αύξηση των πόρων, ούτω ώστε να ενταχθούν στο επόμενο πολιτέ πλαίσιο. Μα είπατε, α, είμαστε ικανοποιημένοι. Μόνο και μόνο από τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν ήδη γίνει. Όχι. Το πραγματικό κίνητρο για να συνεχιστεί θα είναι η πραγματική επιτυχία. Θα την αναλύσετε και θα μα πείτε, για παράδειγμα, ορίστε, εδώ υπάρχει προστιθέμενη εσωτερική αξία. Τότε θα κάνουμε την ουσιώδη συζήτηση, όχι ήδη. Συγγνώμη λοιπόν, εγώ δεν έχω μόνο ποσοτικά κριτήρια, πόσοι έκαναν αίτηση. Θέλω να δω τι διαφορά θα κάνει, τι αλλαγές θα επιφέρει. Σας ευχαριστώ όμως πολύ για τις προσπάθειες που κάνατε. Χαίρομαι που ξεκινάει αυτό το πρόγραμμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πολύ φυσικά θα έχουμε πολύ θετική στάση, θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλλά όχι ακόμη δεν τον είδαμε και για να τον βγάλαμε, Γιατί ε, θα πρέπει να απαντηθούν και αυτές οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ηλικιώτης. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, αρχικά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους εκπρόσωπους της Κομισιόν για την παρουσία και θεωρώ ότι έγινε μια καλή αρχή με την ευκαιρία να ευχαριστήσω ξανά τον εισηγητή από την Επιτροπή μας, τον Κάλλος για τη δουλειά που έγινε και για τη συνεργασία μας. Ω ομάδα τη Ευρωπαϊκή ε, Ενωτική Αριστερά, από την αρχή στηρίξαμε αυτή την πρωτοβουλία για το Wi-Fi. Ε, ωστόσο, για την ομάδα μα, προτεραιότητα είναι να ωφεληθούν από την ασύρματη συνδεσιμότητα ιδιαίτερα τα κράτη και οι περιοχές που είναι λιγότερο ανεπτυγμένες, τα νησιά, οι ορεινές, οι παραμεθόριες, οι απομακρυσμένες και τις πρόσιτες περιοχές. Γιατί ε, μιλούμε για ένα κόστος εδώ ε, και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι πάρα πολλοί ε, δήμοι έχουν την δυνατότητα ε, με δικά τους έξοδα να εγκαταστήσουν αυτή την ασύρματη συνδεσιμότητα. Ε, θα θέλαμε δηλαδή να μας εξηγήσετε επίσης πώς θα διασφαλιστεί ότι ο διαθέσιμος προπολογισμός θα κατανεμηθεί με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο. Ποιε δικλείδε ασφαλεία έχετε ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατόν δημόσιο όφελο και να δοθεί η δυνατότητα στου πολίτε από όλα τα κοινωνικά στρώματα να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα τη συνδεσιμότητα. Αναφέρεται για 4.000 αιτήσει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω από πόσα κράτη-μέλη είναι αυτέ οι αιτήσει. Είναι από όλα τα κράτη-μέλη. Ε, ένα στοιχείο τη πρόταση που μα προβλημάτισε ιδιαίτερα και αυτό το είπαμε πολλέ φορέ και εδώ στην Επιτροπή και κατά τη διάρκεια τη συζήτηση με τον εισηγητή και του άλλου εισηγητέ, είναι ο κανονισμό που πρότεινε η Επιτροπή πόσο προπλεσμό θα κατατίθεται κατά κανόνα με βάση τη σειρά παραλαβής των προτάσεων. First comes, first serve. Για να είναι δίκαιος όμως αυτός ο κανόνας, πρέπει πρώτα να διασφαλιστεί πως όλοι οι υποψήφοι θα έχουν τις ίδιες δυνατότητες για να ανταγωνιστούν. Ε, ποια μέτρα λάβατε λοιπόν ώστε να ενημερωθούν άμεσα τα κράτη και τοπικές αρχές σχετικά με τη σχεδιαζόμενη δράση και τους σχετικούς όρους αλλά και να στηριχτούν επαρκώς γιατί υπάρχουν ε, δήμοι και ε, κοινότητες ε, που δεν έχουν αυτή τα μέσα, αυτή τη δυνατότητα, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τι προεργασίε για την υποβολή των αιτήσεων. Δηλαδή, πόσο λάβαμε υπόψη να βοηθήσουμε ακριβώ κάποιου Δήμου και κοινότητε για να υποβάλουν τι αιτήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Μαρτέν έχει τώρα το Μια ερώτηση έχω πολύ στοιχειώδη. Και εγώ χαίρομαι βέβαια για την πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες κάποια στιγμή να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ε, ψηφιακή ενημέρωση. Αυτό είναι βέβαια θετικό. Ε, έχω όμως μια ερώτηση για τη δημόσια υγεία. Φαντάζομαι ότι χρειάστηκαν επιπλέον κεραίες, εξοπλισμός, οπότε ποιες είναι οι επιπτώσεις των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Έχει γίνει κάποια μελέτη αντικτύπου για την υγεία. Δεν έχει ζητήσει κανείς άλλος το λόγο από ό,τι βλέπω. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον δόκτορα Βιόλα και στον κύριο Γουίλαν και θα ήθελα να πω και εγώ από τη δική μου πλευρά ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα τις προσπάθειές σας αλλά πάντα θέλουμε βελτίωση. Δεν αρκούμαστε σε αυτά που έχουν ήδη γίνει. Εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε στο σωστό θα θέλαμε λοιπόν να μας απαντήσετε στις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω και σε εσά και σε όλους τους ευρωβουλευτές. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά που τέθηκαν οι ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, εισηγητής ο κύριος Ζουρίνιο. Όντως, για μας η υπομονή του και η επιμονή του βρίσκουμε ότι μας βοηθούν πολύ. Φυσικά και εμείς ε, θέλαμε να ξεκινήσει το πρόγραμμα μέσα στην επόμενη μέρα μετά τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα. Όμως ε, τελικά η δημοσίευση που επιτρέπει και την εκταμίευση ήρθε τον Νοέμβριο, παρόλο που σχετική απόφαση είχε ληφθεί τον Ιούνιο. Τι να κάνουμε, αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Το άλλο είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για μία δικτυακή πύλη. Έχουν αναπτυχθεί όλα τα συστήματα τα ψηφιακά για να δοθούν οι επιχορηγήσεις, για να αναγνωριστούν οι δήμοι, για τα κουπόνια κτλ. Δηλαδή, πολλή δουλειά έχει γίνει πάνω σε αυτό ήδη. Καταλαβαίνω την απογοήτευσή του βέβαια. Και εμείς θα θέλαμε σε δύο μήνες να τα έχουμε όλα αλλά είναι αρκετά περίπλοκη η υπόθεση. Τώρα, ποιο είναι το καλό νέο. Το καλό νέο είναι ότι τώρα υπάρχει η πύλη και τώρα μπορούμε να δεχτούμε την εγγραφή πολλών δήμων. Φυσικά, λόγω των περιορισμένων κονδυλίων, θα υπάρχει και περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή δήμων. Αλλά πάντως υπάρχει. δίνουμε 18 μήνες το πολύ. Είναι το ανώτατο όριο, έτσι, για να υλοποιηθεί το Wi-Fi for you. Και για να απαντήσω και στον κύριο Σιλικιώτη, αν ένας Δήμος δεν είναι έτοιμος την πρώτη μέρα, γιατί ίσω δεν γνωρίζουν καλά αυτές τις τεχνολογίες κτλ. Εμεί προσπαθούμε ακριβώ να βοηθήσουμε αυτούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτή την τεχνολογία. Είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον συγκεκριμένο Δήμο για να κάνει τι εγκαταστάσει που χρειάζεται. Αν όμω μπορεί να το κάνει σε μια εβδομάδα, θα το έχει το βάτσο σε μια εβδομάδα. Το λέμε εμεί απλώ για να βοηθήσουμε ακριβώ του Δήμου οι οποίοι αντιμετωπίζουν περισσότερε δυσκολίε με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό, πώς θέλουμε εμείς να λειτουργήσει το σύστημα δηλαδή. Άπαξ έχει εντοπιστεί ο χρήστης και μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε δίκτυο περιαγωγής. Θέλουμε το σύστημα να λειτουργεί με απλό τρόπο. Δεν θέλουμε να προσθέσουμε περιπλοκότητα σε ένα ήδη περίπλοκο σύστημα που θέλουμε να λύσουμε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε πιο περίπλοκο για τους Δήμους. Θέλουμε δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι εφόσον κάποιος έχει εγγραφεί σε ένα τοπικό δήμο, τότε η εγγραφή αυτή μπορεί να ισχύσει και για την εγγραφή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Αυτόματα θα γίνεται λίγο πολύ αυτό. Όχι πλήρως αυτόματο roaming, περιαγωγή, αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι όπως Telecom. Υπάρχουν δηλαδή κάποια τεχνικά στοιχεία που περιορίζουν την κατάσταση. Ε, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε επιπλέον κόστος στους Δήμους. Θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε λοιπόν όλο αυτό το σύστημα Wi-Fi, αλλά να ξέρετε ότι δεν θα πρόκειται για επιπλέον άκθο στους Δήμους. Οι χρήστες όμως θα μπορούν να χρησιμοποιούν το δικό τους ID, όπως λέμε, όνομα χρήστη, και για άλλα δίκτυα. Τώρα για το μέλλον, για το 5G, για να απαντήσω και στον κύριο Μπόνη. Πράγματι, και εδώ απαντάω και στον κύριο Τελίτσικα. ναι, και εμείς είμαστε στραμμένοι στο μέλλον, αυτό κοιτάμε τώρα. Δεν είναι σήμερα η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε τι θα κάνουμε στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι καλώς το Μάιο θα έχουμε την πρόταση της Επιτροπής, όμως έχουμε δει ότι υπάρχει ενδιαφέρον για να πάμε προς την κατεύθυνση χρήσης απλών εργαλείων. Και ναι, βέβαια, σήμερα μας καλέσατε και σας δίνουμε τα στοιχεία που έχουμε τώρα για τις 4.000 εγγραφές ας πούμε. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το πρώτο συμπέρασμα που βγάζουμε το πρώτο 24ωρο ανοίγματο της πύλης είναι ότι υπάρχει ευρεία ζήτηση. Οπότε και εμείς από εδώ, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πρέπει να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε. Κανονικά είναι αρμοδιότητα των περιφερειακών εθνικών αρχών, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτά τα δύο να μην συνδυαστούν μεταξύ τους. Οπότε στο μέλλον, εάν επιπλέον από το Wi-Fi έχετε δυνατότητες 5G και διάφορες κοινότητες όπως είναι τα νοσοκομεία μια άλλοι το χρειάζονται. Ναι, είναι μια δυνατότητα και αυτή προκειμένου να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινότητες περισσότερο. Και ελπίζω επίσης η επιτυχία αυτή να μας επιτρέψει να μιλάμε με διαφορετικούς όρους από εδώ και πέρα με τις χώρες μέλη. Δηλαδή, υπάρχουν χώρες μέλη που έχουν εμπλακεί περισσότερο και άλλες που έχουν αντιταθεί σε αυτή την πρωτοβουλία και ακριβώς από τέτοιες χώρες μέλη έρχονται οι περισσότερες αιτήσει. Οπότε η χώρα η οποία είχε αντιταθεί αρχικά θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Δεν πρέπει να έχουμε αντιστάσεις, αντίθετα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί. Και θα αξιολογήσουμε την εφαρμογή, βεβαίως. Όταν θα έχουν μπει στο σύστημα όλοι οι εγγεγραμμένοι, θα κάνουμε σιγά σιγά την αξιολόγηση. Στην κυρία Γκρίφιν τώρα θέλω να πω ότι είναι. Φυσικά και θέλουμε να βοηθήσουμε με υπηρεσίες, όχι μόνο την υγεία, αλλά και τον τουρισμό και όλα. Και θα υπάρξει αξιολόγηση εξ Θα φροντίσουμε επίσης να υπάρχει αρκετή διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία για όλους προκειμένου να γίνει καλά η αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτού του προγράμματος. Και σε σύγκριση με υπολογισμό ακόμα και της διευκόλυνσης ιδέοντας με την Ευρώπη, αυτό είναι πάρα πολύ μικρό το ποσό. Η επιτυχία πάντως του πρώτου 24ωρου είναι πολύ κατάφορη. Και στον κύριο Τελίτσκα θέλω να πω όχι, εντάξει, δεν έχουμε εξισκωθεί να φωνάζουμε πω πω τι ωραία που πετύχαμε εδώ στο μετρό στις Βρυξέλλες. Όχι, απλώς λέμε ότι δεν ε, περιμέναμε 24 ώρες μετά να έχουμε τόσο πολλές ε, αιτήσει και εγγραφές, 5% των Δήμων δηλαδή να έχουν εγγραφεί ήδη στο πρώτο 24ωρο. Αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν λέω ότι καταλήγω σε συμπεράσματα. Φυσικά και καταλαβαίνουμε ποια είναι τώρα η πρόκληση να κατανείμουμε τα κουπόνια, να βεβαιωθούμε ότι το σύστημα λειτουργεί, ε, πράγμα που σημαίνει ότι οι πρώτοι μήνες θα είναι ιδιαίτερα εντατικοί από πλευρά δουλειά, Και να δούμε βέβαια και τι θα προβλέψει το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Πάντως, ένα, όχι ακριβώ συμπέρασμα, αλλά τέλο πάντων ε, μία εντύπωση είναι ότι πρέπει και εμείς να πούμε στις χώρες μέλη, όχι στο κοινοβούλιο, στις χώρες μέλη που μας είπαν στην αρχή ότι δεν χρειάζονται χρήματα για τα ψηφιακά, τώρα με το 8 δισεκατομμύρια που ήταν η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην αρχή και είπαν όχι, δεν έχουν δίκιο. Αυτοί που είπαν ότι δεν υπάρχει ζήτηση από τους Δήμους και πάλι, να, το αποτέλεσμα τους διαψεύδει. Αυτό που έγινε δηλαδή το τελευταίο 24ωρο. Και αυτοί που είπαν ε, θα δούμε κατά πόσο λειτουργεί το σύστημα, κατά πόσο η κατανομή των vouchers θα γίνει ικανοποιητικά κλπ. Ε, αυτό μένει βέβαια να το αποδείξουμε το ότι θα λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορώ να σας πω ότι αυτό είναι επιτυχία ήδη από σήμερα. Πάντως τα στοιχεία που έχουμε στη θέση μας σήμερα δείχνουν ότι πάει καλά το πράγμα. Και στον κύριο Σιλικιώτη. Τα κοπόνια αυτά είναι για τις κοινότητες που δεν έχουν Wi-Fi. Δηλαδή η κατεύθυνση είναι προς τις κοινότητες εκείνες που είναι λιγότερο προχωρημένες, άρα που είναι λιγότερο στο κέντρο μιας χώρας μέλους. Συγχρόνως, όπως εξήγησε και ο συνάδελφος ο κύριος Βίλαν, θέλουμε να διασφαλίσουμε μια ελάχιστη γεωγραφική κατανομή των κουπονιών στην κάθε χώρα μέλος. Δεν μπορεί κανείς να ελέγξει το κάθε κουπόνι, γιατί τελειώς το σύστημα θα γίνει ιδιαίτερα περίπλοκο. Συζητήθηκε από το Κοινοβούλιο και ήταν μια από τις ευθύς λύσεις που βρήκαμε το, ο πρώτος που κάνει αίτηση είναι ο πρώτος που εξυπηρετεί. Αλλά έχετε δίκιο ότι πρέπει να προβάλλουμε πολύ την προσπάθεια αυτή και να την εξηγήσουμε. Έχουμε σε όλες τις γλώσσες την τεκμηρίωση. Έχουμε ένα help desk. Τι, 100 απευθύνθηκαν σε αυτό χτε, 100 χτες από διάφορους δήμους, σε 24 ώρες δηλαδή. Οπότε υπάρχει το helpdesk για να δίνει απαντήσεις. Και φυσικά θα είναι ένα θέμα. Το ομολογώ. Χτες μπορεί να το σκεφτόμουν διαφορετικά, αλλά ο αριθμός των κουπανιών πράγματι δεν θα φτάσει. Δεν θα ήταν σοβαρό να υποσχεθούμε χρήματα που δεν διαθέτουμε, αλλά θα ήταν σοβαρό να αρχίσουμε να μιλάμε με τις τοπικές αρχές και να προσπαθήσουμε με τις τοπικές αρχές, όπως είπε και ο κύριος Σουρίνιο, τη δυνατότητα μιας εταιρικής σχέσης. Να πούμε δηλαδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δικιά μας υποδομή, τα κουπόνια μας κτλ. Ας συνεργαστούμε αν έχετε και εσείς κονδύλια για να δούμε πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε. Πρέπει να δούμε λοιπόν πρώτον εάν όντως όλα τα κουπόνια θα εξαντληθούν από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει, θα δούμε. Και το δεύτερο βήμα θα είναι να μιλήσουμε με τις εθνικές, με τις τοπικές αρχές και να πούμε, να, ποιες είναι αιτήσει που έχουμε ε, από τη δικιά σας χώρα μέλος, μπορείτε να βοηθήσετε. Και το τρίτο βήμα βέβαια θα είναι στο μέλλον να προβληματιστούμε και σε απόλυτα μαζί σας να έχουμε την κατάλληλη συζήτηση για το νέο προσανατολισμό στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η απάντησή μου στον κύριο Μαρτά είναι απλή. Έχουμε Wi-Fi σε όλα μας τα σπίτια και εδώ, σε αυτό το χώρο. Οπότε, ναι, θα υπάρξει συμμόρφωση με τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτό ναι. Δεν θα μπορούν να εγκατασταθούν εξοπλισμοί τα λοιπά, εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους κανόνες. Και ο εξοπλισμός, ο οποίος θα εγκατασταθεί, προφανώς και θα είναι συμμορφούμενος προς τις διεθνείς προδιαγραφές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι η απάντηση ήταν διεξοδική. Ευχαριστούμε τον ε, δόκτορα Βιόλα, διότι δεν μας έχει συνηθίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τόσο διεξοδικές απαντήσεις. Και έτσι μπορούμε να συνεργαστούμε πολύ καλά και για αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ και ευχαριστούμε τον κύριο Ζωρίνιο και νομίζω ότι θα ξαναβρεθούμε στο εγγύς μέλλον. Μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κανονισμός για τον ΕΝΙΖΑ, Οργανισμό για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο και κατάργηση του προηγούμενου κανονισμού σε σχέση με την πιστοποίηση ασφαλείας στον κυβερνοχώρο. Δίνω το λόγο στην Αγγέλικα Νίμπλερ που είναι και η συγγήτριά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που συζητάμε θέματα κύβερνο ασφάλειας. Καταρχάς, ε, να τονίσω ότι έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Δεν πρόκειται να υποβάλω σχέδιο έκθεσης. Τώρα, γιατί δεν την έχω τελειώσει ακόμη. Θα την τελειώσω μέχρι τέλο τη εβδομάδα και θα τη στείλω στη μετάφραση. Να κάνω καταρχά δύο παρατηρήσει πριν μπω στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, θεωρώ ότι είναι καλό που η Επιτροπή έκανε αυτή την πρόταση. Που έχει μια στρατηγική δηλαδή η Κομισιόν Ασφάλεια, γιατί τα θέματα αυτά εδώ στην Ευρώπη μας ε, απασχολούν εδώ και καιρό. Ξέρετε ότι Υπάρχει ήδη οδηγία για, ε, τα θέματα, για τα συστήματα δικτύων και πληροφορίας που εφαρμόζονται από τα κράτη-μέλη. Συζητάμε ιδιαίτερα τα θέματα στήριξης της ε, ψηφιακής κοινωνίας και του ψηφιακού κλάδου, το 4.0. Αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει μόνο αν υπάρχει εμπιστοσύνη στην ασφαλεία των ε, προϊόντων, των υπηρεσιών και των συστημάτων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μία πρόταση για την ε, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Έχουμε εδώ τα εφή, τους ευφύείς οίκους, τις ευφύείς λύσεις, τις ευφύείς πόλεις. Όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν μόνο αν έχουμε πολύ ψηλό επίπεδο ασφάλειας. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι ασφαλή ότι δεν θα μπορούν να μπουν μέσα hacker, ότι δεν θα υπάρχει κατασκοπία. Και αν διαβάσουμε τι συμβαίνει στον κόσμο, πριν από δύο μέρες έγινε επίθεση hacker στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών και προέκυψε ότι ήταν μια ρωσική ομάδα hacker που λέγεται Βατόλα που μπόρεσε να πάρει και εμπιστευτικά στοιχεία για τις διαπραγματεύσεις για τον Brexit για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία. Δηλαδή στοιχεία που όλα έπρεπε να είναι απόρριτα. Θα ξέρετε την περίπτωση ε, μια συγκεκριμένης ε, κούκλας παιχνιδιού που κατέγραφε όλα όσα γινόντουσαν στα δωμάτια των παιδιών μέχρι που κάποιο του πήρε είδηση στη Γερμανία και αφαιρέθηκε. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Και βλέπετε τι προέκυψε και από τι για την ασφάλεια των τσίπ, των ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Τα υπενθυμίζω. Γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα λοιπόν αυτό που μας απασχολεί και αν δεν επιτύχουμε να έχουμε συστήματα που να διασφαλίζουν την ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών, τότε πολλά από αυτά που θέλουμε να προωθήσουμε δεν θα μπορέσουν να προωθηθούν. Δεύτερον, προκατακτικό. Έχουμε μια ισχυρή βιομηχανία, ένα ισχυρό κλάδο σε όλα τα κράτη-μέλη και άρα με την κυβερνοασφάλεια θα μπορούσαμε να έχουμε και εδώ δηλαδή σε αυτό το τομέα πρωτοπόρο ρόλο. Βεβαίω με βάση και το σωστό νομικό πλαίσιο. Αυτό θέλουμε να διατυπώσουμε. Και ελπίζω ότι θα το επιτύχουμε με αυτή την ε, νέα πράξη. Λοιπόν, να περάσω τώρα στην πρόταση και θα κάνω και μερικές ακόμη παρατηρήσεις. Η πράξη αυτή έχει δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά τον οργανισμό των ΕΝΙΣΑ και το άλλο είναι το σύστημα πιστοποίησης στα κράτη-μέλη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λοιπόν, πρώτον, για τον οργανισμό ΕΝΙΣΑ. Όπως ξέρετε, συνάδελφοι, είναι κατεστημένος ε, στην ε, Αθήνα και το Ηράκλειο. Η ακριβής ονομασία είναι Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και της Πληροφορίας. Από ό,τι ενημερώθηκα, εργάζεται πολύ σωστά, με θαυμάσιους εμπειρογνώμονες που κάνουν πολύ καλή δουλειά και τα παρουσίασε όλα αυτά. Αλλά είναι ένας μικρός φορέας. Έχει 80 εργαζομένους και στο μέλλον θα γίνουν 120. Οπότε το θέμα είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ενίσα. Η Κομισιόν προτείνει να λάβει μια μόνιμη εντολή δηλαδή να έχει και μόνιμο μέλλον. Και προτείνεται να λάβει και περισσότερο προσωπικό και περισσότερη πρικοδότηση. Χαιρετίζω αυτές τις προτάσεις και συμφωνώ. Και ως Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε ακόμη πιο φιλόδοξοι. Δεν αρκεί να πάνε στους 120 εργαζόμενοι. Θα μπορούσαμε να προτείνουμε 500 εργαζόμενους. και υπενθυμίζω πόσους εμπειρογνώμονες έχουν οι εθνικοί οργανισμοί κυβερνοασφάλειας, για παράδειγμα στη χώρα μου, BSC λέγεται σε εμά. έχει 880 εργαζόμενους. Στη Γαλλία είναι πάνω από 500. Αν δούμε και οι εταιρείε ε, τι τμήματα κυβερνοασφάλειας έχουν, από πολλές δεκάδες μέχρι 200 έχουν οι επιχειρήσεις. Γιατί τα θέματα αυτά έχουν πολύ ψηλή προτεραιότητα. Πρώτον αυτό. Διαπιστώνουμε επίσης ότι η ΕΝΙΣΑ λειτουργεί σωστά, πρέπει να αναπτυχθεί, έχει τεράστιο δυναμικό και για να ε, συντονίσει τις εργασίες της, αλλά με βάση τους αριθμούς που σας παρουσίασα, Πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Δεν πρέπει δηλαδή να είμαστε υπερβολικοί. Η ενίσα ξέρετε σαν ένα παιδάκι. Πρέπει να αναπτυχθεί αλλά με ένα λογικό ρυθμό. Και κάνω προτάσεις ε, που θα συνοδεύσουν ακριβώς αυτή τη διαδικασία ανάπτυξης. Δεν θέλουμε να πάρουμε αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη. Κανένας δεν το θέλει αυτό. Αλλά τα κράτη-μέλη θέλουμε να ενισχύσουμε εφόσον θα έχουν και αυτόν τον συμπληρωματικό πυλώνα της ΕΝΗΣΑ που θα έχει αρμοδιότητες περισσότερο για τη λειτουργική συνεργασία. Αυτά τα αναφέρει και η έκθεση. Και το θέμα είναι πόσο θα μπορούσε να συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Όταν θα δείτε το σχέδιο έκθεσής μου, θα τα δείτε πιο αναλυτικά. Λοιπόν, και καταλήγω τώρα για την πιστοποίηση. Κάναμε πολλές ακροάσεις για το θέμα αυτό. Με εμπειρογνώμονες υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα όπου περιμένω και τη δική σας συμβολή. Για παράδειγμα, πρώτα απ' όλα το πεδίο εφαρμογή. Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις από αυτού. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε μόνο τον κύκλο ζωής του κλάδου όταν αναφερόμεθα σε πιστοποίηση. και θα πρέπει οι ορισμοί ε, στους οποίους το βασιστούμε να είναι ευρύς. Αν έχουμε έναν ευρύ ορισμό, θα πρέπει βεβαίως κατόπιν να κάνουμε και μία ιεράρχηση. Γιατί υπάρχουν ε, δισεκατομμύρια μηχανήματα IoT. Δεν είναι δυνατόν να τα πιστοποιήσουμε όλα, θα πρέπει να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες και γι' αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί, να σωστή διαδικασία. Κατά λίγο, αλλά ξέρετε είναι η πρώτη φορά που συζητάμε ένα τόσο σημαντικό θέμα για να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Γι' αυτό σας παρακαλώ ε, λίγη υπομονή, γιατί είναι σημαντικό θέμα. Το δεύτερο θέμα. Εάν θα είναι εθελούσιο ή υποχρεωτικό το σύστημα πιστοποίηση. Εγώ θέλω να βασιστούμε στην εκτίμηση των κινδύνων. Δηλαδή, να, λέμε, να δέμε, ε, ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητα θα είναι ή εθελούσια ή υποχρεωτική πιστοποίηση. Αλλά θα ακούσω με ενδιαφέρον και τι προτάσει των συναδέλφων επ' αυτού. Γιατί υπάρχουν ε, και διαφορετικά επίπεδα ασφαλεία με διαφορετικέ απαιτήσει ανά επίπεδο. Και μπορούμε βεβαίω ε, να έχουμε διαφορετικέ απόψει και για του ορισμού, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικέ αντιλήψει. Θα ακούσω του συναδέλφου. Λοιπόν, πολλά είπα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι και με την ενίσχυση και με την πιστοποίηση να διασφαλίσουμε να έχουμε καλή δομή διακυβέρνηση. Να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία και των κρατών μελών και, η τεχνογνωσία του, και την τεχνογνωσία του κλάδου. Για την πιστοποίηση θα χρειαστούμε και τον κλάδο που αναπτύσσει τα προϊόντα, τα συστήματα, τις, τις ε, υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετάσχει και ο κλάδος. Οπωσδήποτε. Τώρα πώς θα το πετύχουμε αυτό υπάρχουν διαφορετικές ε, δυνατότητες. Θα προτείνω ορισμένα πράγματα και θα ακούσω και τις προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και τους κοιόδης. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, καρποφόρα ανταλλαγή απόψεων. Και βεβαίω θα ακούσω τώρα και αυτά που έχετε να πείτε και μετά θα το ξαναζητήσουμε και όταν θα υποβληθεί η έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Νίμπλερ. Κατανοώ ότι το θέμα ήταν, ε, είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό υπερεύει το ε, χρόνο της. Από τους σοσιαλιστές ο κύριος Κουρουμπασεύ. Ευχαριστώ πολύ. Έχει μεγάλη σημασία να έχουμε χρόνο και για μια συζήτηση σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστούμε την κυρία Νίμπλερ για τις ε, προσπάθειες της. Είναι μια πολύ καλή βάση για συζήτηση με την εισηγήτρια και υπάρχει πολύ θετική ατμόσφαιρα η οποία ελπίζω να επικρατήσει μέχρι τέλους. Ε, υπάρχουν τρία μέρη σε αυτή την πρόταση τα δύο τμήματα αφορούν το ρόλο του ΕΝΙΖΑ και θα θέλαμε να συγχαρούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την πρόταση. Η πρόταση αυτή ενισχύει τον Οργανισμό Ασφάλειας στον κυβέρνοχώρο. Γιατί ε, δεν ήταν πολύ φιλόδοξο το σχέδιο μέχρι τώρα. Νομίζω ότι αν αυξηθεί το προσωπικό από 80 σε 120 θα ήταν καλύτερη η κατάσταση, αλλά τώρα υπάρχουν 80 υπάλληλοι. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε 600 στο γαλλικό οργανισμό, 800 ή 900 στο γερμανικό οργανισμό. Είναι λογικό να υπάρχει α, αυτός ο πολλαπλασιαστικός παράγων επί 12 σε ορισμένα κράτη. Βεβαίως, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δίνουν μεγάλη σημασία στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και πρέπει να τις συγχαρούμε, αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσει και η ασφάλεια του ευρωπαϊκού κυβερνοχώρου, γιατί το ανοιχτό ερώτημα είναι ότι σε περίπτωση κυβερνοεπίθεση σε περισσότερα κράτη-μέλη, ποιος θα αναλάβει μία ενιαία απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή απόκρουση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί πολλές χώρες θα βρεθούν σε δυσχερή θέση. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε το ρόλο του ενίσα ο οργανισμός αυτός ασφάλειας στον κυβερνοχώρο πέρα από την ταυτοποίηση του προβλήματος και της αναφοράς του στην ε, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να προβεί και σε ένα μεγαλύτερο έργο. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε χώρες όπως η Σιγκαπούρη υπάρχει μια συγκεκριμένη υποδομή και σε επίπεδο πρωθυπουργών. Ένας εξοπλισμός. Γι' αυτό τα κράτη-μέλη δεν πρέπει να είναι εγωκεντρικά θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό οργανισμό γιατί πολλές υπηρεσίες δεν θέλουν να ε, ανταλλάξουν πληροφορίες και έτσι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κυβέρνο έγκλημα εκτός και αν γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών ως προς την εθελούσια πιστοποίηση οι εμπλεκόμενοι φορείς θεωρούν ότι θα πρέπει να παραμείνει η εθελούσια βάση, αλλά άλλες χώρες πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης, άρα υποχρεωτικό, όπως γίνεται σε άλλες χώρες και σε άλλες χώρες όπως η ΙΠΑ, η Ινδία και η Κορέα. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τον οργανισμό και στην ανταλλαγή απόψεων ελπίζω να συνεισφέρουμε για την ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της Ευρώπης. Ευχαριστούμε. Ε, το Ζενόφσκι στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Νίμπλερ για τα αρχικά της σχόλια. Πρόκειται για ένα θέμα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία και ενδιαφέρον, γιατί υπάρχουν εγκληματικά κυκλώματα τα οποία επιτίθεται στα δικά μας συστήματα στον κυβερνοχώρο. Και δυστυχώς είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Η κοινωνία πρέπει να είναι σε θέση να μηνθεί. Επιθέσεις σε συστήματα πληροφοριών μπορεί να είναι επιθέσεις απέναντι στην ίδια μας την κοινωνία και την ακυρότητά της. Όπως είπε και η κυρία Μίγκλερ, όσον αφορά τον οργανισμό ΕΝΙΣΑ, συμφωνώ ότι πρέπει να έχουμε έναν ισχυρό οργανισμό και αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή προκειμένου η ΕΝΙΣΑ να αποκτήσει μια μόνιμη εντολή και περισσότερους ανθρώπινους ε, και οικονομικούς πόρους. Κοιτώντας τα έγγραφα πάνω στα οποία εργαζόμαστε, η ΕΝΙΣΑ, η υπηρεσία της ΕΝΙΣΑ, αποκτά όλο και περισσότερες αρμοδιότητες. Πρέπει βέβαια να δουλέψει βάση των δομών που υπάρχουν ήδη στις χώρες μέλη. Κάποιες χώρες μέλη έχουν πολύ ισχυρά συστήματα, οι υπηρεσίες ασφάλειας στο κυβερνοχώρο, άλλες πάλι μόλις τώρα ξεκινούν. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό είναι η αποτελεσματικότητα. Αλλά συγχρόνως να ξέρουμε ότι τα συστήματα που είναι λιγότερο ε, κεντρικά είναι και πιο αποτελεσματικά. Ο ΕΝΙΣΑ λοιπόν δεν θα έπρεπε να είναι με τέτοια δομή κεντρικού χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των επιθέσεων στο κυβερνοχώρο. Δηλαδή αυτό που έχει σημασία είναι να χτίσουμε πάνω στις εμπειρίες που έχουν ήδη οι χώρες μέλη και έτσι να βρούμε καλούς τρόπους συνεργασίας. Κατά τη γνώμη μου, αυτό θα πρέπει να είναι και το κύριο καθήκον του ΕΝΙΣΑ. Το ερώτημα βέβαια είναι σε τι βαθμό ο ΕΝΙΣΑ πρέπει να αναλάβει και λειτουργικές αρμοδιότητες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Πάντως, δεν θα πρέπει, πιστεύω, να αναθέσουμε πάρα πολλές λειτουργικές αρμοδιότητες πάνω στον ΕΝΙΣΑ. Περισσότερο να κατανέμει τις πληροφορίες, να φροντίσει για το συντονισμό μεταξύ χωρών μελών. Τέτοια πράγματα πρέπει να κάνει ο ΕΝΙΣΑ. Έρχομαι τώρα στο θέμα των πιστοποίησεων. Πιστεύω ότι θα είναι περίπλοκο. Έχουμε να κάνουμε εδώ με συμφέροντα διαφόρων κλάδων. Όπως λέει και η κυρία Νίμπλερ, έτσι και εγώ πιστεύω ότι η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται σε θελοντική βάση, κατά κανόνα. και να βασίζεται σε μια ιδιαίτερα λεπτομερή ανάλυση κινδύνου. Αυτή η προσέγγιση που βασίζεται στην ανάλυση κινδύνου δηλαδή λειτουργεί πολύ καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Νότια Κορέα όπου έχουν μεγαλύτερη εμπειρία με αυτά. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία του κλάδου και να χτίσουμε πάνω στις διεθνείς προδιαγραφές. Έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε για να ε, φτιάξουμε και εμείς τις δικές μας ε, προδιαγραφές ασφάλειας. Έχω τη τιμή να συνεργάζομαι με την κυρία ε, Νίμπλερ, έχουμε συνεργαστεί δηλαδή στο παρελθόν για διάφορα ζητήματα. Πιστεύω ότι είναι μια καλή βάση για τη δουλειά μας, η πρότασή της και θα μπορέσουμε έτσι να προωθήσουμε τους στόχους της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα και πρέπει να υποφεληθούμε από αυτή τη στιγμή όσο μπορούμε περισσότερο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τιλτσίκα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στελίτσκα. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Νίμπλερ και τους άλλους συναδέρφους για τα όσα είπαν. Καλά τα περιέγραψαν, υπάρχουν διάφορες διαστάσεις στην ασφάλεια στον κυβερνό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλά κενά και σε μερικά πράγματα έχουμε μείνει πίσω, υπάρχει κάποια δράνεια. Η διάσταση των καταναλωτών είναι πολύ σημαντική και ξέρουμε πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί αν πληγεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Τώρα το μέγα ζήτημα εδώ δεν είναι τόσο ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε εμείς εδώ στην Ήτρια για το θέμα. Το θέμα είναι τι λένε οι πολιτικοί στις χώρες μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι πρόβλημα νοοτροπία μερικές φορές. Σε κάποιες χώρε μέλη, συγγνώμη για αν υπερβάλλω εδώ κάπως, αλλά ορισμένοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Και εμεί θα είμαστε τόσο δυνατοί όσο δυνατός είναι ο πιο αδύναμος κρίκος τη αλυσίδα. Συνεπώ αυτό το οποίο εδώ χρειαζόμαστε οπωσδήποτε είναι σημαντική αλλαγή τη νοοτροπία. Και έτσι να καταλήξουμε σε ένα ρυθμιστικό περιβάλλον που θα αναβαθμίσει τα πιο αδύναμα τμήματα της αλυσίδας. Αυτή ήταν η πρώτη παρατήρηση. Τώρα, ο Ενίσα, αναφερθήκαμε στον οργανισμό αυτό, κάνει καλή δουλειά κατά τη γνώμη μου. Κρίνοντας από τις ανοιχτές πηγές, δεν ε, είχα πολλές ευκαιρίες. Μίλησα δύο φορές στην Ελλάδα με τον διευθυντή και όντως αντιμετωπίζουν τα ζητήματα πολύ ρεαλιστικά για τους στόχους τους. Όμως το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ είναι ότι παρόλο που θα ήταν πολύ καλό να έχουμε ένα κανονισμό ο οποίος να ισχύει επιμακρό και να μας οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της κυβερνοασφάλειας, αυτό δεν γίνεται γιατί ο κόσμος αλλάζει και κάθε τρία-τέσσερα χρόνια ε, θα έχουμε αλλαγές και οι κίνδυνοι θα είναι διαφορετικοί. και από την άλλη στο Συμβούλιο όλο και περισσότεροι θα θέλουν να καταλήξουν στο επίπεδο ασφάλειας που θέλουμε κι εμείς. Οπότε ίσως θα έπρεπε εδώ πέρα να προχωρήσουμε σταδιακά και να εξηγήσουμε ποιο θέλουμε να είναι το επόμενο βήμα με κάποιες ρήτρε ασφαλείας, ότι θέλουμε ένα στέρεο σύστημα με συνεχή βελτίωση της ασφάλειας εννοείται ότι και εγώ είμαι υπέρ μιας μόνιμης εντολής και ενίσχυσης του ενίσα. Τώρα σε τι επίπεδο δεν ξέρω, γιατί εξαρτάται και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει όταν αποφασίσουμε ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του ενίσα. Να επικεντρωθούμε στα εξή θέματα. Σε εθελοντική βάση όχι. Το Συμβούλιο τι θα κάνει πρώτο. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να ξεκινήσουμε με την εθελοντική βάση και θα δούμε μετά. Αλλά από την άλλη, αν είναι σε εθελοντική βάση, τι γίνεται με τη βιωσιμότητα. Εμείς τι ομάδα στοχεύουμε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκτενώς ή όχι θα χωρίσουμε θέματα στρατηγικής σημασίας. Πρέπει να δούμε τι επίπεδο θέλουμε. Και ξέρετε ότι μπορείτε και μέσα από μια τηλεόραση να χακάρετε το σύστημα ή το, με το ρολόι των παιδιών σας. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πάντως ένα ζήτημα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι πώς θα δώσουμε θετικά κίνητρα. Γιατί από πλευρά του καταναλωτή, αν δει ότι κάτι έχει ευρωπαϊκό σήμα και το σήμα αυτό το δίνει ο ΕΝΙΣΑ, αν είναι κάτι το οποίο προβλέπει κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές, τότε έχω και περισσότερο εμπιστοσύνη ότι μπορώ με ασφάλεια να αγοράσω αυτό το προϊόν. Άρα να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ρύθμιση από τη μια και από την άλλη μεριά σε κάτι το οποίο θα επιτρέψει αυτορύθμιση και καλύτερη συνειδητοποίηση του καταναλωτή. Και θα τελειώσω με το εξή. Διάφορα ζητήματα πρέπει να εξετάσουμε και σίγουρα δεν είναι εύκολο. Πρέπει να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Και σας είπα ήδη μερικά, ίσως το ένα τρίτο από αυτά που θα ήθελα να εξετάσουμε και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε καλές διατάξεις. Θα μπορούσα να συνεχίσω επί μακρό, αλλά αυτή είναι ο πρώτος προσανατολισμός, η πρώτη συζήτηση σήμερα. Ευχαριστώ. Mm, ο κύριος Νταλούντε από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια για αυτό το σχέδιο, η ΟΕΝΙΣΑ θα μπορέσει πραγματικά να είναι ένας παράγων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, εάν έχουμε τη σωστή οικοδόμηση, καταρχήν σταθερότητα. Εάν δεν υπάρχει εντολή, τότε δεν θα έχουμε να κάνουμε με έναν μόνιμο εταίρο. Επίσης, να υπάρχει ανταπόκριση στους, στις προκλήσεις του τομέα καθώς και εφαρμογή της ασφάλειας με σχεδιασμό και ιδιωτικότητας. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει μία απλή και διαφανής διαδικασία και τέλος και εξίσου σημαντικό το πλαίσιο πιστοποίησης θα πρέπει να προβάλλει ε, ε, ένα σχέδιο το οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε μέσα στα πλαίσια της αγοράς και να μην έχουμε θέση σε εμπορία προϊόντων όπου υπάρχουν κίνδυνοι ανασφάλειας. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία αν λάβουμε υπόψη την, ε, τις ε, γρήγορες εξελίξεις του τομέα. Σε σχέση με την εθελούσια πιστοποίηση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σημεία εισόδου τα οποία όμως να μην έχουν έλλειψη προδιαγραφών ασφάλειας. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν εξοπλισμός ο οποίος ε, δεν έχει μια διαδικασία εισόδου με password και είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα και θα το κάνουμε μέσω των τροπολογιών μας. Ευχαριστούμε πολύ γιατί ήσασταν και ιδιαίτερα σύντομος. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ματίας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή τη στιγμή το θέμα της ασφάλειας του κυβερνοχώρου είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε ότι δυστυχώς γίνονται κυβερνοεπιθέσεις με συγχωρείτε, σε πολλά κράτη-μέλη. Είδαμε τι έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με φορολογικούς ε, ε, παραδείσους, αλλά έχει σχέση με την Cambridge Analytica, η οποία χρησιμοποίησε προσωπικά δεδομένα έτσι ώστε να επηρεάσει εθνικές εκλογές. Κάτι το οποίο δεν είχαμε δει στο παρελθόν. Πρόκειται για ένα παιχνίδι, ένα παιχνίδι που το χρησιμοποιούν όλοι με βάση συγκεκριμένες εφαρμογές και το Facebook. Άρα υπάρχει θέμα ιδιωτικότητας και αυτό το σκάνδαλο φύγει αυτό το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό το είδαμε και με βάση τις αποκαλύψεις του Σνόντεν. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτά τα σχήματα εξαπάτησης που επηρεάζουν ακόμα και εθνικές εκλογές. Δεν είναι ένα θέμα που αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά θέμα ελευθερίας και δημοκρατικών διαδικασιών. Νομίζω ότι θα πρέπει να συγχαρούμε την εργασία των δημοσιογράφων γιατί συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα που αφορά την ελευθερία της ε, δημοσιογραφίας και το μέλλον της. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα ζητήματα ε, είναι στο επίκεντρο της καθημερινότητάς μας και αυτό αφορά και το πώς πλήττονται οι πολίτες. Δεν μιλάμε για αφηρημένα αφηγήματα όπως υπηρεσίες και εξοπλισμός. Νομίζω λοιπόν ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σημαντική, αλλά είναι κενή περιεχομένου επί της ουσίας. Δεν ανταποκρίνεται σε τέτοια ζητήματα. Επίσης, επικρατεί σύγχυση σε αυτή την ανακοίνωση. Μιλάμε για θέματα του ΕΝΙΖΑ, της εντολής του, του προσωπικού και από την άλλη μιλάμε για την ευρωπαϊκή πιστοποίηση για την ασφάλεια στον χώρο. Ως προς τον ΕΝΙΖΑ νομίζω ότι θα πρέπει να απαντήσουμε τάχιστα και συντονισμένα στις κυβερνοεπιθέσεις στον ευρωπαϊκό χώρο και γι' αυτό ο ΕΝΙΖΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συνδράμει τα κράτη-μέλη για να ανταποκριθούν σε τέτοιες επιθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει όμως να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί δεν πρέπει να πληγεί η ιδιωτικότητα και οι δημοκρατικές διαδικασίες. Ως προς την πιστοποίηση είναι απολύτως απαραίτητη και ο ΕΝΙΖΑ θα πρέπει να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και όχι μόνο με μερικούς και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει ο απότερος στόχος να είναι η προστασία των καταναλωτών. Όταν μιλάμε για υποχρεωτική ή εθελούσια πιστοποίηση θα πρέπει να ξέρουμε για τι προϊόντα μιλάμε. Ίσως θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική πιστοποίηση για τα πιο ευαίσθητα προϊόντα και εξοπλισμούς. Είναι πολύ δύσκολο το έργο της κυρίας Νίμπλερ και θα προσπαθήσουμε να συνδράμουμε σε αυτό το έργο έληξαν και οι παρεμβάσεις των σκιωδών. Τώρα θα παρέμβουν άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να είναι σύντομοι. Μπόνι. Thank you very much, for Ευχαριστώ, Αγγέλικα. Πολύ καλή παρουσίαση δεν μας περιέγραψες αυτό το πακέτο απλώς, αλλά μας ε, έθεσες και κάποιες εναλλακτικέ επί των οποίων πρέπει να τοποθετηθούμε. Πρώτον, πρέπει να ενισχυθεί η ενίσα, πολύ σημαντικό. Διότι μόνο η ενίσα μπορεί να διασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Επίσης, πρέπει να τη στηρίξουμε και να δημιουργηθεί ένα νέο πρότυπο ανταλλαγής πληροφοριών όταν έχουμε επεισόδια, για να μαθαίνουμε όταν γίνονται επιθέσεις. Χρειαζόμαστε ένα τέτοιο οργανισμό στην Ένωση και για αναλυτικά θέματα. Για να αναλύσουμε, για παράδειγμα, τους κινδύνους και οι λύσεις να βασίζονται σε αποτίμηση των κινδύνων και η ΕΝΙΣΑ θα μπορέσει να συλλέξει στοιχεία και να προτείνει λύσεις. Δεύτερον, τα προγράμματα πιστοποίησης. Συμφωνώ ότι δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι για να εισαγάγουμε υποχρεωτικά τέτοια συστήματα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια εθελούσια πιστοποίηση και να δώσουμε την προοπτική του, του υποχρεωτικού. Γιατί ξέρετε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει πιστοποίηση. Θα πρέπει να λειτουργούν με βάση την αγορά. Βεβαίως δεν έχουμε μία λύση για όλα τα προβλήματα. και επίσης θα πρέπει να βελτιωθεί και η κατανόηση από πλευράς του κοινού των θεμάτων κυβερνοασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ. Μπλάνκο Λόπεθ. Ευχαριστώ. Ορισμένες φορές όταν συζητάμε για ευρωπαϊκούς οργανισμούς αντιμετωπίζουμε κάποιους που είναι αρνητικοί έναντι οποιοδήποτε προϋπολογισμού ε, οργανισμών. Αλλά αυτό το θέμα είναι ζωτική σημασία για του πολίτες. Κάθε μέρα ακούμε ειδήσει για επιθέσεις κυβερνοασφάλεια σε, στις πιο διαφορετικές υπηρεσίες τις οποίες ε, εκμεταλλεύονται για διάφορους σκοπούς. Το τελευταίο πολύ σοβαρό παράδειγμα είναι αυτή η ιστορία του Facebook. Η Ευρώπη πρέπει να έχει τα αναγκαία μέσα για να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τις κυβερνοεπιθέσεις ιδιαίτερα όταν είναι θέματα τόσο σημαντικά όπως η ηλεκτρονική υγεία, τα διασυνδεδεμένα οχήματα και οτιδήποτε έχει να κάνει με το ίντερνετ των πραγμάτων, διότι τα προβλήματα ασφαλείας αυτού του τομείς μπορεί να στοιχήσουν ζωές. Αλλά βέβαια πρέπει να είναι οι λύσεις ανάλογα με τα προβλήματα, που να μπορούν να προβλέψουν και καταστάσεις του μέλλοντος σε έναν τομέα που έχει τρομερή τεχνική πολυπλοκότητα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πρόταση οδεύει προς σωστή κατεύθυνση. Ε, όχι, οδεύει προς σωστό στόχο. Ευχαριστώ πολύ. Πιλάρ Δελκαστήλιο. Ευχαριστώ. Χθε το βράδυ η κυρία Νίμπλερ και εγώ συμμετείχαμε σε μια συζήτηση όπου υπόθηκε ότι η κυβερνοασφάλεια θα είναι ένα από τα θέματα τα πιο σημαντικά της τελευταίας δεκαετίας. Όχι. Δεν είναι σωστή η διατύπωση αυτή. Η κυβερνοασφάλεια θα είναι το σημαντικότερο θέμα για την υπόλοιπη ζωή μας, όπως η ασφάλεια γενικά είναι μόνιμα με πρώτη προτεραιότητα. Συμφωνώ με πολλά που υπόθηκαν. Για παράδειγμα, πρέπει να διευρυνθεί η εντολή, να δοθούν περισσότεροι πόροι στον οργανισμό αυτό ενίσα, συμφωνώ. Θεωρώ να, ότι είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε από πού θα ξεκινήσουμε. Διότι ξέρετε ότι στον επιγραμμικό κόσμο οι κανονισμοί πάντα υστερούν της πραγματικότητας και ο κίνδυνος είναι ότι θα καθυστερούν έτη φωτός από την πραγματικότητα. Θα πέχουν. Πρέπει λοιπόν και για την πιστοποίηση να κάνουμε περισσότερα και κυρίως να καθορίσουμε τις σωστές προτεραιότητες. Να μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς βέβαια υπερβολική ρύθμιση. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τέτοιες ρυθμίσεις ακόμη και σε επίπεδο ενό κράτου μέλους είναι δύσκολες, Άρα σε ενωσιακό πολύ χειρότερες. Πρέπει να υπάρχει σωστή σχέση μεταξύ ιεράρχηση, ελαστικότητας, ευελιξίας. Όλα αυτά πρέπει από κοινού να τα συμφωνήσουμε. Η κυβερνοασφάλεια θα είναι το σημαντικότερο θέμα που θα απασχολήσει τις κοινωνίες, τις κοινωνίες μας από εδώ και στο εξή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δύο είναι τα ερωτήματα και πολύ καλά τα έθεσε η κυρία Νίμπλερ. Ποιο είναι το αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας και ποιος είναι ο ρόλος του οργανισμού ΕΝΙΣΑ. Το αποδεκτό επίπεδο ασφάλειας πρώτα απ' όλα. Υπενθυμίζω, άκουσα τις προτάσεις, τις τοποθετήσεις των συναδέρφων που λένε καλύτερα σε θελοντική βάση και όχι υποχρεωτικά. Ναι, αλλά γιατί όχι, λέω εγώ. Αν δεν υπάρχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει υποχρέωση από τι χώρε μέλη για πιστοποίηση, δεν θα υποχρεώσουμε ούτε καν τι χώρε μέλη να συνεργαστούν μεταξύ του. Γιατί δεν υπάρχει λόγο χώρες οι οποίες έχουν ιδιαίτερα ψηλό επίπεδο όπω η Γαλλία, η Γερμανία, που έχουν όντω πολλούς εκατοντάδες επιρογνώμονες και εργαστήρια πιστοποιημένα που δουλεύουν και κάνουν δοκιμέ σε πραγματικά μεγέθη, γιατί θα συνεργαστούν. Μιλάμε σήμερα, μιλήσαμε πριν από λίγο για το Wi-Fi για όλους. Και μετά λέμε να μείνει σε θελοντική βάση αυτό. Μα όχι, ο κόσμος είναι συνδεδεμένος μεταξύ του και οι επιθέσεις όντως θα υπάρχουν περισσότερες. Εσείς το είπατε, δεν υπάρχει μικρή ή μεγάλη ασφάλεια, υπάρχει ένα επίπεδο που πρέπει να επιβάλλουμε για να μπορέσουμε να είμαστε προστατευμένοι. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε και να καθησυχάσουμε τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές. Εγώ πριν από δύο μήνες η τράπεζά μου μου είπαν ότι κάποιοι χακάραν τον αριθμό του λογαριασμού μου και προσπάθησαν στην Μπαγκόκ να βγάλουν χρήματα από το δικό μου το λογαριασμό. Κάποιος δηλαδή είχε χακάρει τα δικά μου τα δεδομένα, αλλά το σύστημα ασφάλειας ήταν αποτελεσματικό και αυτοί που προσπάθησαν να, ε, να πετύχουν κάτι δεν το πέτυχαν. Οπότε σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να έχουμε τις καλύτερες προδιαφέσεις ασφάλειας. Υποχρεωτικά. Και αλλιώς δεν τα καταφέρουμε. Μην ξεχνάμε τι γίνεται στις ΗΠΑ και στην Κίνα που έχουν συστήματα πιστοποίησης, χειρότερα από τα δικά μας, πιο χαμηλά, και να ξέρετε ότι οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι θα κερδίσουν κομμάτια της αγοράς μας για την κυβέρνηση ασφάλεια. Και εμείς θα χάσουμε και τα συμβόλαια αλλά και την ασφαλειά μας. Γι' αυτό λοιπόν η συνεργασία και το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των χωρών μελών θα εξαρτηθεί από το επίπεδο ασφάλειας που θα ζητήσουμε. Και γι' αυτό πρέπει να ενισχυθεί και ο ΕΝΙΣΑ. Λοιπόν, να δούμε ποιε είναι οι πραγματικέ λειτουργίε, η αποστολή τη ΕΝΙΣΑ και ανάλογα με αυτό που θα του ζητήσουμε να κάνουν, να αποφασίσουμε και για τα μέσα. Εγώ δεν λέω πόσα, αν είναι 150, 200 ή 1000, δεν ξέρω. Εξαρτάται από το ρόλο του ενίσα. Αν χρειάζεται χίλιους, να έχει χίλιους ανθρώπους. Είναι στρατηγική επιλογή αυτή. Αλλιώς, τίποτα δεν θα κάνει η ενίσα. Ξεχάστε το. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστούμε που δίνετε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια για την πρότασή μας. Έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις από ό,τι ακούμε. Οπότε αυτό που έχει τώρα νόημα είναι να δούμε πού υπάρχει σύγκληση με το Συμβούλιο για την πρόταση όσον αφορά τον οργανισμό ΕΝΙΣΑ. Υπάρχει σύγκληση ε, ανάμεσα σε αυτά που λέτε εσείς δηλαδή εδώ σήμερα και τις χώρες μέλη, που σημαίνει ναι, μόνιμη εντολή και πιο ισχυρό οργανισμό. Ρωτάτε κατά πόσο οι πόροι και με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρκούν προκειμένου να παίξει το ρόλο της ο ΕΝΙΣΑ. Και αυτό συνδέεται βέβαια και με τα καθήκοντα του οργανισμού τηρίζεται ο ρόλος του ΕΝΙΣΑ όσον αφορά τόσα κάνει μέχρι τώρα, αλλά το ζήτημα στο Συμβούλιο είναι ο ρόλος του ΕΝΙΣΑ όσον αφορά την πιστοποίηση. Και αυτό είναι κάτι που και εσείς το είπατε. Αν υπάρξει κρίση, επίσης ποιος θα είναι ο ρόλος του ΕΝΙΣΑ. Εμείς θέλουμε ένα συμπληρωματικό ρόλο με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για να μην υπάρχει επικάλυψη με αυτά που κάνουν οι εθνικοί αντίστοιχοι οργανισμοί. Οπότε και η πρότασή μας δεν έχει σαν στόχο την επικάλυψη. Καθ' άλλο. Προσθέτει στα όσα ήδη υπάρχουν στην οδηγία. Όπως ξέρετε, ο ΕΝΙΣΑ έχει ως ρόλο συνεργασία με τα εθνικά δίκτυα. Οπότε ίσως χρειάζεται εδώ κάποια διευκρίνηση. Πάντως φάνηκε εδώ ότι υπάρχει στήριξη από εσά. Για την πιστοποίηση αυτή καθ' αυτή. Πράγματι, συμφωνούν και οι χώρες μέλη. Γίνεται συζήτηση για την ανάλυση κινδύνου, για διαφάνεια στο σύστημα. Κατά πόσο πρέπει να υπάρχει τώρα αυτοπιστοποίηση ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο συζητούν οι χώρες μέλη. Η Επιτροπή προτείνει την εθελοντική βάση. Αυτό σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στο πρόγραμμα δεσμεύεται για την εποπτεία και την εφαρμογή του συστήματος. Αυτό είναι ένα σύστημα αυτορύθμισης που δεν υπήρχε στον κανονισμό πριν. Και για την υποχρέωση πιστοποίησης, την υποχρεωτική δηλαδή πιστοποίηση, θέλω να αναφερθώ σε αυτό που είπε ο κύριο Τελίτσκα, δηλαδή να, γίνει, να υπάρχει μια προσέγγιση βήμα-βήμα. Έχουμε ήδη τη βάση προκειμένου προγράμματα να γίνουν υποχρεωτικά σε κάποιου τομείς. Στο άρθρο 47, για παράδειγμα, εξηγούμε ότι το πρόγραμμα πιστοποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσφέρει ακριβώς την πιστοποίηση ασφάλειας προκειμένου να τηρηθεί η αρχή της καλύτερης ρύθμισης. Θέλω να πω ότι ήδη υπάρχει δυνατότητα κάποια προγράμματα να γίνουν υποχρεωτικά και να καλύπτονται κάποιοι τομείς υποχρεωτικά. Τώρα γιατί δεν το προτείναμε ως ε, κομισιόν είναι γιατί ακόμα δεν υπάρχει βεβαιότητα για το εύρος εφαρμογής και το πόσο μακριά πρέπει να πάμε. Αυτό που κάναμε είναι ότι δημιουργήσαμε διαφορετικά επίπεδα διασφάλισης που θα επιτρέψουν στην αγορά να αποφασίσει. Όσον αφορά τη συμμετοχή των χωρών μελών. Και εδώ στο Συμβούλιο γίνονται συζητήσεις. Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, οι χώρες μέλη έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν προτείνοντας ευρωπαϊκά προγράμματα πιστοποίησης. Συνεπώς, προτείνουμε να δημιουργηθεί μια ομάδα ευρωπαϊκής πιστοποίησης που να προτείνει προγράμματα πιστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί το κάνουμε έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε το όλο θέμα. Κάποια αναφέρθηκαν στις αρμοδιότητες του ΕΝΙΣΑ. Ο ΕΝΙΣΑ πράγματι, όπως είπε κάποιος, είναι ένα μωρό που μεγαλώνει. Τώρα κάνει πολλή δουλειά για την ασφάλεια, αλλά πρέπει να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και να ενισχυθεί. Το να του αναθίσουμε διάφορα επιπλέον καθήκοντα πιστοποίησης θα είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να διαχειριστεί. Τώρα, στην πρόταση της Επιτροπής προβλέπεται ο ΕΝΙΣΑ να ζητεί γνωμοδότηση από τους διάφορους εταίρους και φορείς σχετικά με την πιστοποίηση. Ίσως και εδώ χρειάζεται διευκρίνηση και γίνεται συζήτηση στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο προχωράει πολύ καλά λοιπόν, όπως γνωρίζετε και εμείς είμαστε στη διάθεση της Επιτροπής σας για να σας βοηθήσουμε. Πολλές φορές μας έχετε δώσει την ευκαιρία να έρθουμε και να συζητήσουμε μαζί σας για αυτά τα θέματα, οπότε είμαστε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την εισήγηση και νομίζω ότι αυτό το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά. Η κυρία Νίμπλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για αυτά τα σχόλια. Αυτές οι πρώτες ε, εκτιμήσεις είναι πολύ καλές. Μιλάμε για πιστοποίηση σε εθελούσια ή μη βάση. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριστεί, γιατί τη στιγμή που υπάρχουν προϊόντα στην αγορά λειτουργούν πολύ καλύτερα σε θελούσια βάση. Αλλά φυσικά θα πρέπει να υπάρχει μια βάση ασφάλειας και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την διαφοροποίηση των προϊόντων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και θα σας μιλήσω για την τελική έκβαση της έκθεσης. 24 Απριλίου του 2018 θα μπορούμε να δούμε την έκθεση συνολικά μετά τις τροπολογίες. Περνάμε στο επόμενο θέμα που αφορά την ενημέρωση της αποστολής της, ε, ε, Επιτροπής στην Χιλή με έξι μέλη που βρέθηκαν στη Χιλή από τις 18 μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λεβαντόφσκι, ο οποίος θα ήθελα να λάβει υπόψη και το χρόνο, τα χρονικά πλαίσια, γιατί θα έχουμε και την παρουσία του Επιτρόπου αργότερα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για αυτή την αποστολή. Μιλήσαμε για τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας με τη Χιλή, συμφωνία σύνδεσης με την Χιλή και χρειάζεται χρειάστηκε μεγάλη συνδρομή και από την άλλη πλευρά ήρθαμε σε επαφή με τον ε, ε, Υπουργό Ενέργειας, τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων. Είδαμε, επισκεφθήκαμε το Κογκρέσο και τη Γερουσία και ήρθαμε σε επαφή και με την Ένωση του Ειρηνικού και της Καραϊβικής. Αυτό που είχε μεγάλη σημασία για μας ήταν το παρατηρητήριο με τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια που προσελκύουν τους περισσότερους επιστήμονες από όλο τον κόσμο και αυτή η ε, επίσκεψη ήταν πολύ σημαντική. Η Χιλή είναι μια σταθερή χώρα από πολιτικής και οικονομικής πλευράς. Είμαστε βεβαίως σε άμεσο ανταγωνισμό με την Κίνα και την Ιαπωνία για να έχουμε εμπορικές σχέσεις με την Χιλή και στον τομέα της αιωλικής και ηλιακής ενέργειας μπορούμε να βοηθήσουμε στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, της επιστήμης και θα πρέπει να αναβαθμίσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί για ιστορικούς λόγους θεωρούν την ευρωπαϊκή συνεργασία Ω συνεργασία με την Ιβυρική Χερσόνησο για ιστορικούς καθαρά λόγους. Ε, υπήρχε καλό έτσι συλλογικό πνεύμα συνεργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες. Ωραία. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λεβαντόφσκι και περνάμε στο επόμενο θέμα που αφορά την αποστολή στη Γενέβη 19-21 ε, Δεκεμβρίου για την συμμετοχή στο Φόρουμ για την διακυβέρνηση του διαδικτύου. Η συνάδελφος έχει το λόγο. Thank you very much. Προς τον συνάδελφο, ο συνάδελφος Μπόνι έχει το λόγο. Όπως ξέρετε, το 2017 ε, το Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου, το IGF, διοργανώθηκε στη Γενέβη και εγώ ήμουν επικεφαλής της δικής μας αντιπροσωπείας, ε, του Κοινοβουλίου δηλαδή, σε συνεργασία με την Επίτροπο Μαρία Γκάμπριελ, η οποία ήταν και πρόεδρος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επίτροπης. Είχαμε συναντήσεις με νέους σε σχέση με το μέλλον του διαδικτύου και επίσης εστιάσαμε την προσοχή μας στην ασφάλεια, στην ε, ε, προστασία της ιδιωτικότητας και στην αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων. Είχαμε και άλλες χώρες από το γειτονικό χώρο και ήρθαμε σε επαφή και με πολλές ε, ΜΚΟ, α, ε, ε, οργανώσεις των πολιτών και μιλήσαμε για την ελευθερία του διαδικτύου, γιατί όταν μιλάμε για ορισμένα ζητήματα στη Λατινική Αμερική ή την Αφρική, η κατάσταση φαίνεται εντελώς διαφορετική από τη δική μας ευρωπαϊκή οπτική. Προβήκαμε σε ανταλλαγή απόψεων ήταν καρποφόρα η συνεργασία και για εκείνους και για εμάς. Μιλήσαμε και με εκπροσώπους του επιχειρηματικού χώρου, γιατί κατέστη σαφές ότι κατά τη συνάντηση αυτού του φόρουμ μας ενδιαφέρει και ο μελλοντικός σχεδιασμός του διαδικτύου Μιλήσαμε για την αγορά εργασίας στο μέλλον και πώς ε, ε, το εργατικό δυναμικό θα μπορέσει να, θα πρέπει να προσαρμοστεί όταν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα αναπτυχθεί και θα συνεργάζεται με το ανθρώπινο δυναμικό. Συζητήσαμε και για το θέμα της ουδετερότητας του διαδικτύου και ήταν, ε, όπως ξέρετε, μεγάλη σημασία αυτό το θέμα εξαιτίας της τάσης των ΙΠΑ. Μιλήσαμε και για το 5G. Θέλουμε να κατέχουμε ηγετική θέση, αλλά και η Νότια ωραία. μας μίλησε για τις πρώτες εμπειρίες με 5G κατά τους, κατά τους Ολυμπιακούς, χειμερινούς Ολυμπιακούς και αυτό αφορά και την Ιαπωνία η οποία θα προβάλλει αυτή την ταχύτητα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Επίσης, συνεργαστήκαμε και με το ευρωπαϊκό IGF, το οποίο θα συνέλθει στην Τυφλίδα. Εάν θέλετε λοιπόν, μπορείτε να λάβουμε υπόψη την ανάπτυξη αυτού του συστήματος, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολύ κοντά. Θα καλέσουμε εκπροσώπους από τις Βαλκανικές χώρες και από τη Βόρειο Αφρική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, συζητήσαμε μετά το φόρουμ, το IGF, για κάτι κρίσιμο σε σχέση με τα πρότυπα δηλαδή του φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Τώρα θα πρέπει να δούμε το Eurotic που είναι το ευρωπαϊκό IGF για τις επιχειρήσεις, για την κοινωνία των πολιτών σε σχέση με ψηφιακά ζητήματα για το μέλλον. Και αυτή είναι η πρώτη χρονιά, το 2018, όπου δεν γνωρίζουμε ε, που θα λάβει χώρα το IGF, που θα συνεδριάσει αυτό το φόρουμ. Μάλλον στο Βερολίνο, του, για του χρόνου τουλάχιστον, το 2019, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το φετινό IGF. Γι' αυτό καταβάλουμε προσπάθειες για να υποστηρίξουμε το φόρουμ στην Τυφλίδα. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μπόνι, άκρος ενδιαφέροντα όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ε, παρεμβάσεις από τους ε, συμμετέχοντες. Και τώρα θα ε, ασχοληθούμε με την αποστολή στην Αυστρία. Δεν είναι εδώ όμως ο κύριος Ρούμπιχ εδώ Γι' αυτό θα ασχοληθούμε με το επόμενο θέμα για την ενημέρωση σχετικά με τις ε, διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, όλα τα θέματα είναι πολύ σημαντικά αυτά που μας απασχολούν και αυτό είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες. Τελευταία φορά που μας απασχόλησε ήταν το 2009, δηλαδή σχεδόν πριν από μία δεκαετία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει τόσο εντυπωσιακά που η κατάσταση να είναι εντελώ διαφορετική. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε τα δίκτυά μας και τις υποδοσμές μας για τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας προηγμένης ψηφιακής οικονομίας, να εξυπηρετεί την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να ανταποκρίνεται και στην προηγμένη ψηφιακή κοινωνία. Βεβαίω λοιπόν μας απασχολεί ο ανταγωνισμός, η προστασία των καταναλωτών, όπως πάντα. Αλλά ο κύριος στόχος μας αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε ένα αριθμιστικό πλαίσιο που θα ενισχύσει τις υψηλές επενδύσεις που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε 500-600 εκατομμύρια για να έχουμε ένα δίκτυο υψηλής ε, αποδοτικότητας ε, οπτικών ινών για να έχουμε τις, ε, την εφαρμογή της τεχνολογίας 5G. Η οδηγία λοιπόν αυτή έχει δύο κύρια στατικά που είναι η ουσία του ζητήματος. Από την μία έχουμε το φάσμα. Είχαμε δυσχέρεια στο καθορισμό μιας ευρωπαϊκής πολιτικής διαχείρισης του φάσματος. Διότι τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι το φάσμα ήταν θέμα επικουρικότητας. Πολύ απρόθυμα. Θα θυμάστε και σε άλλα νομοθετήματα που περάσαμε πρόσφατα για την ουδετερότητα κτλ. Ενώ το φάσμα ε, ήταν τμήμα της συζήτησης, δεν δέχτηκε το Συμβούλιο να συζητηθεί λέγοντας όχι, όχι, δεν θα μας απασχολήσει. Τώρα λοιπόν καταλήγουμε σε αυτόν τον κώδικα. όπου το φάσμα είναι ζωτικό τμήμα. Αλλά άλλαξε η κατάσταση. Γιατί οι εξελίξεις τα τελευταία 2-3 χρόνια των ψηφιακών τεχνολογιών είναι τόσο σοβαρές που διαπερνά παντού την οικονομία. Άρα χρειάζονται παντού οι καλύτερες υποδομές από πλευράς ταχύτητας, ποιότητας, και τα λοιπά. Τι μπορούμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε καταλήξαμε σε συμφωνία, γιατί τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα. Αλλά υπάρχει κάποια συμφωνία για το φάσμα που μπορούμε να πούμε ότι είναι επιτυχία για το Κοινοβούλιο. Γιατί έχουμε ασκήσει τόση πίεση για να υπάρξει ένα κοινό πλαίσιο για την διαχείριση του φάσματος. Ενώ παλιά δεν είχαμε καμία πολιτική γι' αυτό και θα διαμορφωθεί μια κατάσταση που θα ισχύσει για 20 ετία, τουλάχιστον 20 ετία για τη χρήση του φάσματος, για το δικαίωμα χρήσης. Άρα είναι πιο ελκυστικό για τους επενδυτές. Επίσης ε, υπάρχει ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι όμως ε, εντάσσονται σωστά στο πλαίσιο αυτό το γενικό, το εξυπηρετούν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες κοινοί κανόνες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προσελκύσουν λοιπόν και αυτοί οι επενδυτές. Και κάτι καινούριο που προέκυψε από τη συζήτηση. Είπαμε και συμφωνήσαμε ότι πριν από το 2020 η, η τα διαστήματα συχνοτήτων που έχουν να κάνουν με την εισαγωγή του 5G θα πρέπει να έχουν αποφασιστεί. Για το 5G λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σίγουρα τις κατάλληλες ε, υποδομές από πλευράς φάσματος. Τώρα λοιπόν συζητάμε τα θέματα πρόσβασης στα δίκτυα. Θέλουμε λοιπόν και εδώ να έχουμε ρυθμίσεις που θα προωθήσουν τις επενδύσεις. Τα, τα συζητάμε λοιπόν τώρα στο Συμβούλιο και με τη συμμετοχή της Επιτροπής βεβαίως ε, ως ε, διαμεσολαβητού. Καλά τα πάμε από πλευρά ρυθμού, Βέβαια απέχουν ε, ορισμένες θέσεις του Συμβουλίου από τις θέσεις του Κοινοβουλίου, αλλά έχουμε μια θαυμάσια ομάδα. Όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι σκιώδες είναι εξαιρετικοί. Ε, είναι ο κύριος Τοζανόφσκι, ξέρει πως πάντα πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι τα πάμε καλά και θα επιτύχουμε καλή συμφωνία και για τα θέματα πρόσβασης. Θα δούμε τι θα γίνει στον επόμενο βέβαια τριμερή διάλογο, αν θα μπορέσουμε να κλείσουμε όλα τα ανοιχτά θέματα, γιατί υπάρχουν και μερικά ακόμη που εκκρεμούν. Οπότε, με βάση την πείρα μου, νομίζω ότι είναι ένας από τους καλύτερους τριμερείς διαλόγους από όσους έχω συμμετάσχει. Σας ευχαριστώ λοιπόν, ευχαριστώ το προσωπικό μας και τους συνεργάτες ε, των βουλευτών και τους υπαλλήλους της Ήτρε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Θα δώσω το λόγο για αυτό το μέρος της ενημέρωσης, γιατί άλλοι δεν είναι παρόντες σε σχέση με, τον, ε, ενεργειακό, με, την ενεργεια, με τις ανανεώσιμες ενέργειες, ε, μπλανκολόπες, ενεργειακή απόδοση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υπάρχει επικύρωση. Ε, στήριξη Επιτροπή μας και ολόκληρο το Κοινοβούλιο την θέση μας όσον αφορά τις ανανεώσιμες ενέργειες. Κάτι το οποίο μας έδωσε μεγάλη ενέργεια για να μπούμε στις διαπραγματεύσεις. Είχαμε ένα τριμερή διάλογο μέχρι τώρα, ο οποίος ήταν εισαγωγικό. Δηλαδή το κάθε δυσμικό όργανο εξήγησε την τοποθέτησή του και έθεσε έτσι τις βάσεις για την διαπραγμάτευση των συμβιβασμών. Διαπιστώσαμε σε αυτήν την πρώτη συνάντηση ότι οι θέσεις Συμβουλίου και Κοινοβουλίου βρίσκονται μακριά εμένα από τις ΔΕ σε διάφορα ζητήματα όπως είναι η θυμιστική ασφάλεια, η μεταφορά, ε, η αυτοκατανάλωση και άλλα. Υπάρχουν όμως και θέματα με τα οποία συμφωνούμε. Έγιναν διάφορες τεχνικές συναντήσεις με στόχο να τεθούν οι οι κατευθυντήριε γραμμέ τέλο πάντων για να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις και να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα σεβασμό του τριμερεί διαλόγου. Ο επόμενος είναι στις 27 του μηνό. Η Προεδρία πάντως θα φέρει σύντομα μία εντολή για να συζητήσουμε σε βάθος και έτσι να δούμε τι συμφωνία μπορούμε να πετύχουμε. Κατά τη γνώμη μου η Βουλγαρική Προεδρία κάνει καλή δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα της Προεδρίας για την αφοσίασή της, για τη σκληρή της δουλειά, αλλά όπως σας είπα, οι διαφορές μεταξύ μας είναι ακόμα μεγάλες, ημών και του Συμβουλίου. Και αυτό παρά τα νέα στοιχεία που έχουν μπει στο τραπέζι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προσπαθεί να λάβει υπόψη του και το Συμβούλιο και εμείς τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών, που είναι από το 2014 και μετά για το κόστος και άλλα, αλλά δεν αλλάζει τη θέση του το Συμβούλιο. Και αυτό αρχίζει να μας ανησυχεί. Όπως σας είπα, ακόμα είμαστε στην αρχή. Εξερευνούμε το πεδίο και ελπίζουμε το Συμβούλιο να πάψει να είναι αδιάλακτο όσον αφορά τη χρήση των ανανεώσιμων ενεργειών να επιτρέψει στους πολίτες τη μετάβαση στην ανανεώσιμη ενέργεια και να έχουμε νέες προτάσεις. Επαναλαμβάνω, είμαστε στην εξερεύνηση των διαφόρων θέσεων και ελπίζουμε στον επόμενο τριμερή διάλογο να έχουμε περισσότερο περιεχόμενο. Επαναλαμβάνω ότι εκτιμούμε όλους ιδιαίτερο το έργο της Βουλγαρικής Προεδρίας γιατί δείχνει ότι ενδιαφέρεται μέσα στην εντολή της να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Όμως, μας μένει πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε. Είμαστε σε αυτό το πρώτο στάδιο, όπως σας είπα, και οι διαφορές μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου είναι ακόμα μεγάλες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο. Ε, είμαστε πεπισμένοι ότι ότι το θέμα βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια. Νομίζω ότι πριν μιλήσουμε για τις δύο τελικές ενημερώσεις, να μιλήσουμε για την αποστολή της Επιτροπής Ήτρε στην Αυστρία 14 με 16 Φεβρουαρίου και θα δώσω λόγο στον κύριο Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι φτάσαμε την κατάλληλη στιγμή. Βεβαίω δεν ασχολήθηκε με την ε, Αυστριακή Προεδρία που θα γίνει το επόμενο εξάμεινο, που θα είναι το επόμενο εξάμεινο. Ούτε ασχολήθηκε με το πολιτές πλαίσιο, ούτε με το Brexit. Κυρίως ασχοληθήκαμε με δικά μας θέματα. Ο Σίτρα, όπου ήταν ο Βέρνα Λάγκε, και ο Θέοντρος Τολογιάν και ο Φλάβιο Τζάνονάτο. Ήταν επίσης και οι κυρίες ε, Μίλναρ και Κάπελ. Και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με το Αυστριακό Κοινοβούλιο. Γιατί διαπιστώσαμε ότι ζούμε σε δύο διαφορετικούς ε, κόσμους. Και είναι καλό λοιπόν να ανταλλάσσουμε απόψεις και να ακούμε τι προβλήματα υπάρχουν. και οι συνάδελφοι του Αυστριακού Κοινοβουλίου είχαν πολύ θετική αντιμετώπιση και τόνισαν ότι θα ήθελαν να μπορούν να κάνουν συχνά τέτοιους αναλυτικούς διαλόγους. Πήγαμε στο στούτο για την κβαντική μηχανική και την οπτική στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών και εδώ ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα προγράμματα έρευνας Ευρωπαϊκής Ένωσης η κυρία Καστίγιο αναφέρθηκε μόλις τώρα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και συζητήσαμε τα θέματα που θα απασχολήσουν τον τομέα αυτό, οι κβαντικές τεχνολογίες. Είναι κάτι που θα μπορούσε να επιφέρει ριζικές ανατροπές ε, σε ολόκληρο το ίντερνετ. Αν υπάρξουν σημαντικές ε, αλλαγές εδώ, σημαντικά επιτεύγματα, μπορεί να προκαλέσει ριζικές αλλαγές παντού. Δηλαδή η ψηφιακή λειτουργία θα είναι πολύ διαφορετική. Επίσης πήγαμε σε μια ε, μεγάλη εταιρεία που ασχολείται όχι μόνο με επιχειρήσεις και προγράμματα στην Ευρώπη, αλλά και στον κόσμο. Πήγαμε σε ένα δηληστήριο και σε ένα κέντρο καινοτομία. και πήγαμε και στον κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου στο Baumgarten. Ε, αποκτά κανείς μια εντύπωση για το τι όγκοι φυσικού αερίου μετακινούνται και τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν. Στο Baumgarten υπάρχουν πέντε εγκαταστάσεις πίεσης ε, 50 μέτρων βάθους. Είδαμε λοιπόν πώς ε, αποθηκεύεται το φυσικό αέριο, πώς μεταφέρεται, πώς διασφαλίζεται δηλαδή η ασφάλεια παροχής. Μετά πήγαμε στο αυστριακό ηλεκτρικό δίκτυο. Είδαμε πώς παράγεται από τη μία ο ηλεκτρισμός και μετά είδαμε πώς μεταφέρεται. Πήγαμε στην ομάδα Continental Euro Το δίκτυο στην Αυστρία έχει 3.400 χιλιόμετρα καλωδίων με 34 σταθμούς υψηλής ε, τάσης Μας υπόθηκε ότι για ορισμένε διαδικασίες χρειάζονται υπερβολικές, ε, υπερβολικά χρονοβόρες ε, περνάει πολλοί χρόνο για να δεθούν κάποιες εγκρίσει. Και τονίσαμε ότι θα ήταν σκόπιμο για κάποια τέτοια σημαντικά προγράμματα, εάν δεν υπάρχουν αντίθετες δικαστικέ αποφάσεις, να θεωρηθεί ότι εγκρίνονται αυτομάτω. Θα θέλαμε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για να προωθήσουμε τις ε, ανανεώσιμες ενέργειες χωρίς τις καθυστερήσεις για περισσότερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Να υπάρχουν αναγκαίες υποδομές, ούτως ώστε στο μέλλον να μπορούμε να παράσχουμε αυτές τις υπηρεσίες στους συμπολίτε μας. Ακούσαμε ότι για να ε, λειτουργήσουν κάτι τέτοια χρειάζεται κανείς ένα φορτηγό πιστοποίησης και εγκρίσης δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει με τόση γραφειοκρατία ο τομέας της ενέργειας. Συζητήσαμε με τον επικεφαλής ενός μεγάλου αυστριακού ομίλου που έχει 400 εργαζομένους όπου συζητήσαμε θέματα επιστημονικής έρευνας, πώς βλέπουν το πρόγραμμα πλαίσιο 9 σε σχέση με την ενέργεια και μας είπαν ότι πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί στον τομέα αυτό. Ήταν πολύ καλή συζήτηση. Την τελευταία μέρα συναντηθήκαμε με την Υπουργό για τα ψηφιακά θέματα, για την ψηφιακή οικονομία και τις μικρομεσαίες. Την κυρία Μαργαρέτε Σφράμπεκ, που προέρχεται από τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και είναι αρμόδια και για το εμπόριο. Είναι αρμόδια για το λογισμικό στην ψηφιακή ενία αγορά και για προγράμματα κατάρτισης. Νομίζω ότι αξιοποιήσαμε κάθε λεπτό της συζήτησης και μάλιστα δεν μας έφτασε ο χρόνος. Κατόπιν πήγαμε στο Υπουργείο Ενέργειας όπου μας είδε ο Δόκτωρ Λος, ο οποίος είναι διευθυντής ο οποίος μας παρουσίασε τις προτεραιότητες του χειμερινού πακέτου, την ε, αποδοτικότητα της ε, ανανεώσιμες και την ε, ασφάλεια της παροχής. Η Αυστρία νομίζω απέδειξε ότι στον τομέα των ανανεωσίμων έχει σημειώσει και θα μπορούσε να σημειώσει ακόμη περισσότερες πρόοδους. Η κυβέρνηση θέλει μέχρι το 2030 να έχει 100% ανανεώσιμες. συναρπαστικό να δούμε πώς το επιτύχει. Μετά πήγαμε στον Υπουργό για εκπαίδευση, έρευνα και τις επιστήμες. Μας είπε ότι θα στηρίξει το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο, να καθοριστεί πριν από τις ευρωεκλογέ. Η Αυστριακή Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί, ούτως ώστε το ένα το πρόγραμμα πλαίσιο να έχει εγκριθεί πριν τις εκλογές. Για μας αυτό θα είναι μια απόδειξη ότι επιτυχάνουμε αυτά που θέλουμε για να μπορούμε να τα πούμε και στο εκλογικό σώμα. Και μετά επισκεφθήκαμε και ένα πολύ ενδιαφέρον κέντρο κατάρτισης αιωλικής ενέργειας που νομίζω ότι είναι ε, πολύ καλό να μαθαίνουν και οι νέοι για τι επιτυχάνει η Ευρώπη για το τομέα της ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενημέρωση. Τώρα έχουμε άλλες τρεις ενημερώσεις για τις διαπραγματεύσεις. Ε, την πρώτη θα την κάνω εγώ, αλλά θα δώσω το λόγο στους Τούρμς και Ριβαζή για το θέμα της διακυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτό το θέμα της διακυβέρνησης. Είχαμε τον πρώτο τρίμερη στις 21 Φεβρουαρίου 18 όπου είχαμε τις αντίστοιχες θέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αν και συζητήθηκε το περιεχόμενο πολλών άρθρων, αλλά δεν λήφθησαν ε, αποφάσεις μαζί με τον συνεισηγητή, τον κύριο Τούρμες, ε, θεωρήσαμε ότι το Κοινοβούλιο έχει μία πολύ εύρωστη εντολή γιατί υποστηρίχθηκε από την Ολομέλεια. Λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν τις μακροχρόνιες στρατηγικές για να τεθούν σε εφαρμογή οι συμφωνίες των Παρισίων καθώς και η στρατηγική απομάκρυνσης από τον άνθρακα και χρήση μεθανίου καθώς και τις προτεραιότητες και την ενεργειακή αποδοτικότητα καθώς και τον μηχανισμό πλήρωσης των κενών. Ε, λήφθησαν υπόψη και οι θέσεις του κυρίου Στανκόφ, του αναπληρωτή Υπουργού Ενέργειας, ο οποίος τόνισε τις ομοιότητες μεταξύ των δύο θέσεων όσον αφορά τις ανανεώσιμες. Ο κύριος Κανιέτε, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ε, προέβη σε μία διαμεσολάβηση ε, έτσι ώστε να δούμε τι θα κάνουμε και με το μηχανισμό της πλήρωσης των κενών. Όσον αφορά το μεθάνιο, η Επιτροπή θα προβεί σε μία έρευνα. Ε, μετά τον πρώτο τριμερή έγιναν δύο τεχνικές συνεδριάσεις όπου συζητήθηκαν πολλά ε, άρθρα στα οποία εδόθη τελική μορφή και έχουν προβλεφθεί και άλλες συναντήσεις. Ο δεύτερος τριμερής θα γίνει την 5η στις 26 Μαρτίου και όλα βαίνουν καλώς γενικά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο συνάδελφος Τούρμες θέλει να προσθέσει κάτι. Νομίζω ότι κινούμαστε πολύ καλά σε τεχνικό επίπεδο, αλλά η θέση του Συμβουλίου είναι πολύ αδύναμη και θεωρούμε ότι γίνεται μια κίνηση από το Συμβούλιο από προοδευτικά κράτη-μέλη, χρειάζονται χρόνο και νομίζω ότι επόμενος τριμερής στα τέλη Απριλίου θα είναι πιο αποδοτικός εάν έχουμε επιτύχει τάχιστη πρόοδο. Εν πάση περιπτώσει έχουμε μια ευρύτατη εντολή από το Κοινοβούλιο. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε ως προς τις φιλοδοξίες μας και τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων. Θα πρέπει να λάβουμε θέση μάχης και θα τη δώσουμε αυτή τη μάχη. Ωραία, σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Το ίδιο μας είπε και ο συνάδελφος Λόπες Μπλάνκο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Λοιπόν, η κυρία Γκροστέτ θα λάβει το λόγο για την βιομηχανική ανάπτυξη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο πρώτος τριμερής έγινε ήδη σε σχέση με την βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας στις 15 Μαρτίου στο Στρασβούργο και φυσικά παρουσίασα την εντολή του Κοινοβουλίου και συνόδευσα τους δύο συναδέλφους από την ΑΦΕΤ, ε, Εστεβαν Κονσάλες Πόνς και Ιωάνν Πάσκου από την ΑΦΕΤ και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Μαζί με την Βουλγαρική Προεδρία θέλαμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις για να τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο κανονισμός την 1η Πρώτου 19, έτσι ώστε να υπάρχουν και οι γραμμές του προϋπολογισμού, οι εγγραφές των προϋπολογισμών, άρα θα πρέπει να τελειώσουμε τις εργασίες τέλη Μαΐου. Δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο. Κατά την πρώτη συζήτηση υπήρξε θέμα ε, προϋπολογισμού των επιλέξιμων και μη οντοτήτων. Εδώ αποκλίνουν οι θέσεις μας, διότι το Κοινοβούλιο δεν θέλει να γίνει η επαναχρησιμοποίηση προγραμμάτων. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το δημοσιονομικό πλαίσιο που δεν έχει αποδοθεί. Το Συμβούλιο θέλει το αντίθετο γιατί εάν υπάρχουν ε, περιθώρια, μάλλον ποσά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, τότε επιστρέφονται στα κράτη-μέλη. Ζητήσαμε από την Επιτροπή να μας προτείνει ένα συμβασμό γιατί θα πρέπει να εξευρεθεί. Δεν μπορούμε να, μείνουμε, να παραμείνουμε σε αυτές τις αποκλίνουσες απόψεις. Θα θέλαμε λοιπόν η Επιτροπή να φτάσει σε ένα συμβασμό που θα γίνει αποδεκτός και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ως προς τις ε, μη επιλέξιμες ε, δράσεις, εκεί προχωρήσαμε. Υπάρχει μία ιδιαίτερη ρήτρα ως προς ε, ορισμένα όπλα που κατασκευάζονται δυνάμει αυτού του προγράμματος και με βάση τις διεθνείς υποχρεώσεις. Εδώ θα υπάρξει συμφωνία. Ως προς το πρόγραμμα εργασίας το Κοινοβούλιο ζήτησε να υπάρχει μια κατεξιοδότηση πράξη γιατί η Επιτροπή θέλει εκτελεστική πράξη. Για μας όμως μία τέτοια εκτελεστική πράξη δεν αιτιολογείται, δεν δικαιολογείται. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τα προνόμια του Κοινοβουλίου έτσι ώστε η βασική πράξη να εμπεριέχει όλες τις ε, βασικές διατάξεις. Εμείς ζητήσαμε εκτελεστική πράξη, διότι το πρόγραμμα δράσης ε, της Επιτροπής δεν διέπεται από ακρίβεια και τη στιγμή που δεν το έχουμε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό το εξήγησα και επέμεινα ως προς τις επιλέξιμες οντότητες και δράσεις πρότεινα περισσότερη ακρίβεια έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά που ε, τις κατέχουν τρίτες χώρες θα είναι επιλέξιμες εάν τηρούνται οι όροι το Συμβούλιο ε, διακατέχεται από μεγαλύτερη αμέλεια, ενώ εμείς είμαστε σταθεροί και αμετάκλητοι. Στις 10 Απριλίου προβλέπεται ο επόμενος τριμερής, θα πρέπει να κινηθούμε τάχιστα, θα γίνουν και τεχνικές συνεδριάσεις, αλλά θα πρέπει να κινηθούμε πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να υποχωρήσει και το Συμβούλιο και η Επιτροπή να υποβάλει αποδεκτές προτάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Διεξοδική και αυτή η παρουσίαση. Έχουμε την ε, εισήγηση για την ενεργειακή απόδοση του κυρίου Πώς. Ο πρώτος ε, τριμερής έγινε στις 22 Φεβρουαρίου, μετά έγιναν τέσσερις τεχνικές συνεδριάσεις όπου επιτελέστη σημαντική πρόοδος για την ε, πρόταση συμβασμού. Μιλάμε για την τιμολόγηση της θέρμανσης και ζεστό νερό για οικιακή χρήση. Επίσης, λάβαμε υπόψη την αρχή πρώτα η ενεργειακή απόδοση και χτες έγινε ο δεύτερος τριμερής. Δεν φτάσαμε σε άλλες αποφάσεις σε σχέση με τα δύο σημεία, δηλαδή μετρήσεις και τιμολόγηση της κατανάλωσης. Χρειάζεται μεγαλύτερη πρόοδος στα άλλα δύο σημεία ε, σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια και το ε, Energy First. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερη απόδοση, ενεργειακή απόδοση και εμείς προβάλλουμε δέσμευση 35% ενώ το Συμβούλιο 30% ως προς την ενεργειακή απόδοση. Επίσης θα πρέπει να γίνει εξοικονόμηση της ενέργειας δυνάμη του άρθρου 7. Εμείς ε, ζητήσει, μάλλον η Προεδρία ζήτησε να γίνει η επόμενη συνάντηση, είχε ε, προτείνει να γίνει στις 13 Μαρτίου, αλλά στη, θα γίνει τελικά τον Απρίλιο στη Σόφια, στις 16 Απριλίου, για να μιλήσουμε για τους τρεις ε, φακέλους που άπτονται της ενέργειας. Στο άτυπο συμβούλιο η Προεδρία θα μπορέσει να προβάλλει μία συμφωνία συμβασμού και θεωρούμε ότι θα λήξουν οι διαπραγματεύσεις μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Πόκε και ευχαριστούμε εσάς που μείνατε εδώ μέχρι τώρα. Στις 5 ακριβώς, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο, τον κύριο Σέκοβιτς, σε σχέση με το φυσικό αέριο. Θα σας παρακαλούσα να παραμείνετε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη διακοπή ολίγων λεπτών. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, τώρα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μάρο Σεφκοβίτς, Αντιπρόεδρο, αρμόδιο για την Ενεργειακή Ένωση. Αντιπρόεδρο πρώτα απ' όλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι, και πρόεδρο της Ενεργειακής Ένωσης. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι πρόεδρος της Νερική Ένωσης και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μας ενημερώσει σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τον εφουδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Πρώτα απ' όλα, κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ξέρουμε ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, αρχές Μαρτίου, όταν η Προμγκάζ αρνήθηκε να εφοδιάσει την Ουκρανία με ήδη προπληρωμένο φυσικό αέριο και θέλει μάλιστα να αποσυρθεί από τη σχετική σύμβαση. Και μάλιστα μια εποχή που οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα χαμηλές. Οπότε και οι κρανικές αρχές έπρεπε να πάρουν έκτακτα μέτρα και να κλείσουν κάποιες διευκολύνσεις. Μην ξεχνάμε ότι το 2006 και ιδιαίτερα το 2009 η κατάσταση ήταν πολύ παρόμοια στην Σλοβακία και στη Βουλγαρία. Δεν υπήρχε φοδιασμός φυσικού αερίου για δύο εβδομάδες και μάλιστα στο βαθύ χειμώνα. Οπότε γνωρίζουμε τι σημαίνει αυτό. Τώρα λοιπόν είχαμε μια αντίστοιχη κατάσταση στην Ουκρανία. Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε τον κύριο Αντιπρόεδρο, να του ζητήσουμε μάλλον να μας εξηγήσει λιγάκι το πολιτικό πλαίσιο και τις εξελίξεις όσον αφορά αυτό το θέμα, ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, για την ασφάλεια εφοδιασμού ε, φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μέτρα θα πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή μάλλον έχει ήδη πάρει προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Θα θέλαμε να τα ξέρουμε αυτά ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή μας που είναι και πιο αρμόδια για το όλο ζήτημα. Οπότε και πάλι ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Έχετε και το λόγο κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ αξιότιμε Πρόεδρε, αγαπητέ Ζέρση, αξιότιμε Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε να ανταλλάξω απόψεις με την Επιτροπή σας Ήτρα όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον φοδιασμό της Ουκρανίας με ρωσικό φυσικό αέριο. Η Επιτροπή σας, ε, το γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι ασχολείται όλος ιδιαίτερος με το όλο περίπλοκο ζήτημα της Ενεργειακής Ένωσης. Και αυτό γιατί η ενεργειακή ασφάλεια και οι εξωτερικές επιτυχίες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και ξέρω ότι αυτά τα θέματα σας απασχολούν πολύ, σας ενδιαφέρουν πολύ. Και είναι τιμή για μένα που είχα την ευκαιρία πολλές φορές μέχρι σήμερα να έρθω και να τα συζητήσω μαζί σας. Πιστεύω ότι ακριβώ χάρη σε αυτές τις επαφές μεταξύ μας καταφέραμε μαζί να καταλήξουμε σε σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα έλεγα ότι αποτελούν το ακρογωνιαίο λίθο της αρχιτεκτονικής μας για την ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε εγκρίνει νέο κανονισμό για την ασφάλεια εφοδιασμού φυσικού αερίου που επιτρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις εμπορικές συμβάσεις. Και το θυμάμαι πολύ καλά ότι οι χώρες μέλη έλεγαν ότι ποτέ δεν θα συμβεί αυτό. Κι όμως πετύχαμε σημαντικά αποτελέσματα και χάρη στον κανονισμό αυτό μπορέσαμε να θεσπίσουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης κινδύνων. Κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει στην περίπτωση κρίσεων. Εγκρίναμε επίσης την απόφαση για συμφωνιών για το φυσικό αέριο βάσει τις οποίες οι χώρες μέλη διαπραγματεύονται συμφωνίε μόνον εφόσον αυτές συνάδουν με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και θέλω επίσης εδώ να υπογραμμίσω και το δικό σας έργο όσον αφορά τη στατική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το υγροποιημένο φυσικό αέριο που επιτρέπει να διαφοροποιήσουμε το ενεργειακό μας τοπίο. Και ήδη φαίνεται πως οι νέοι σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου έχουν σαν αποτέλεσμα να πέσει η τιμή και επίσης υπάρχουν και νέες δυνατότητες για χώρες που προηγουμένως εξαρτώταν κυρίως από μία πηγή. Υπάρχει τεράστια διαφορά τώρα όσον αφορά το ενεργειακό τοπίο και την ασφαλειά μας για τον ενεργειακό εφοδιασμό. Μαζί λοιπόν δουλέψαμε πάνω σε όλα αυτά και φέραμε και αποτελέσματα όσον αφορά τις υποδομές της ασφαλείας μας. Θέλω εδώ να αναφερθώ ως ιδιαιτέρως στους ε, αγωγούς διασύνδεσης. Ο κατάλογος είναι μακρύς. Έχουμε φροντίσει για αυτούς τους αγωγούς διασύνδεσης που πρέπει να έχουν την ικανότητα εκείνη η οποία μας επιτρέπει, την ικανότητα αποθήκευσης δηλαδή, που μας ε, επιτρέπει να νιώθουμε περισσότερο ασφαλείς. Θα μπορούσα να παριθμίσω πολλά ακόμα μέτρα σχετικά με την αποθήκευση αλλά και άλλα βήματα που έχουμε αναλάβει τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, σήμερα νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι χάρη στη συνεργασία μας και το εξαιρετικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από πλευράς ενεργειακής ασφάλειας σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια. Και αυτό αποδεικνύει ότι η Ενεργειακή Ένωση αποφέρει καρπούς. Στα πλαίσια τώρα της Συμφωνίας των Παρισίων και των στόχων μας για το 2030, επίσης έχουμε ξεκινήσει ανεπιστρεπτή στο δρόμο για ενέργεια χωρίς άνθρακα. Αυτή η μετάβαση της Ευρώπης είναι πλέον ένα γεγονός. Παρ' όλα αυτά, όμως, συγχρόνως, πρέπει να πούμε ότι μέσω πρόθεσμα, ακόμα και αν πετύχουμε τους στόχους μας, το φυσικό αέριο θα παραμείνει σημαντική ενεργειακή πηγή για την Ευρώπη. Χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία για τις ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού σε φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ο λόγος που είναι αυτό τόσο σημαντικό είναι ότι τώρα τα δύο τρίτα περίπου του φυσικού αερίου που καταναλώνουμε στην Ευρώπη εισάγεται από το εξωτερικό. Και βλέπουμε ότι μειώνεται η εσωτερική παραγωγή, άρα η εισαγωγή φυσικού αερίου θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Και εδώ είναι ακριβώς το ζήτημα που παρεμβαίνει με τον εφοδιασμό ρωσικού φυσικού αερίου γιατί συνολικά από τις ε, μη ευρωπαϊκές ε, εισαγωγές είναι περίπου 40% το ρωσικό φυσικό αέριο. Συνεπώς οι σχέσεις μας με την ε, Ρωσία είναι πολύ σημαντικές. Και πριν από λίγο καιρό το είχα πει ότι δουλεύουμε για την ενεργειακή μας ασφάλεια. Θέλουμε να μειώσουμε την εξάρτησή μας και να μειώσουμε την ε, διάσταση του πόσο ευάλωτοι είμαστε σε περίπτωση που κάτι συμβεί στο εξωτερικό. Πρέπει να μπορούμε να συνεχίζουμε να τροφοδοτούμε τις οικονομίες μας. Η Ουκρανία τώρα είναι ένας ε, στενός εταίρος μας, στρατηγικής σημασίας και η Ουκρανία γετονεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ξέρετε έχω υπογράψει ένα νέο μνημόνιο κατανόησης για την ενέργεια το 2016 με την Ουκρανία που θέτει τους όρους για την συνεργασία γύρω από τις πέντε διαστάσεις της ε, Ενεργειακής Ένωσης. Η ενεργειακή συνεργασία πρέπει να βοηθήσει την Ουκρανία να εξυγχρονίσει την οικονομία της, δεδομένου ότι η ενέργεια αποτελεί και δυσποδηλική στήλη της οικονομίας της Ουκρανίας και είναι πολύ βασικό στοιχείο για την σταθεροποίησή της. Η Ουκρανία λοιπόν έχει ξεκινήσει ενεργειακές μεταρρυθμίσεις και έχει ήδη πετύχει πολλά. Είτε πρόκειται για το φυσικό αέριο, είτε πρόκειται για άλλα μέτρα που αφορούν την ενεργειακή επάρκεια. Εμείς βοηθούμε την Ουκρανία όχι μόνο με know αλλά και με οικονομική στήριξη πάνω από 100 εκατομμύρια φέτος, για παράδειγμα. Συγχρόνως, η Ουκρανία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο διότι αποτελεί τη διαδρομή μέσω της οποίας φτάνει το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Ο κύριος Μπούζεκ ήδη αναφέρθηκε στα έτη 2006 και 2009 και μας ε, υπενθύμησε την τραγική κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε όταν διακόπηκε ο αφοδιασμός αυτός. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι που μετά το 2009 και παρά τις γνωστές προκλήσεις στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, η διαδρομή αυτή της Ουκρανίας λειτουργήσε καλά όλα αυτά τα χρόνια. Και χάρη σε αυτήν τη διαδρομή είχαμε αξιόπιστο εφοδιασμό φυσικού αερίου στην Ευρώπη, κάτι το οποίο βέβαια βοηθάει γιατί έτσι τροφοδοτούνται οι οικονομίες μας. Συγχρόνως όμως η μεταφορά αυτή δημιουργεί και έσοδα για την ίδια την Ουκρανία. Και ξέρετε πόσο αναγκαία είναι τα έσοδα αυτά προκειμένου η Ουκρανία να χρηματοδοτήσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι τόσο πολύ σημαντικές για το μέλλον των Ουκρανών. Οπότε δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η ένταση μεταξύ των δύο χωρών που είχαμε τα τελευταία χρόνια με την παράνομη ρωσική κατάληψη της Κρυμαίας και τη φοβερή σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία, πώς λοιπόν η ένταση αυτή επηρεάζει την ενεργειακή κατάσταση τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε πολύ καλά και το τι έγινε με τη διαδικασία διατησίας της Στοκχόλμη. Οι περιπτώσεις διατησίας της Στοκχόλμης, όπως γνωρίζετε, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο σχετικά με τις σχέσεις των δύο εταιριών της, Ναυτογκάς και της ΚΑΣΠΡΟΜ. Τώρα να υπενθυμίσω ότι επιλέγει το δικαστήριο αυτό η διατησία δηλαδή της Στοχόλμης και από τις δύο πλευρές ε, της σύμβασης προκειμένου αυτή η διετησία να ισχύσει στις εμπορικές του σχέσεις. Τώρα δεν χρειάζεται να σας πω τις λεπτομέρειες όσον αφορά την ε, διετησία αυτή και τι ακριβώς έγινε και ποια είναι η διαδικασία. Πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, καλωσορίζει το γεγονός ότι κατέληξε η διατησία της ε, Στοκχόλμης σε μία απόφαση όσον αφορά την ε, μεταφορά του φυσικού αερίου βάσει της σύμβασης Ναυτογκάς με Γκάσπρομ. Και η Επιτροπή περιμένει και οι δύο πλευρές να τηρήσουν τώρα την απόφαση αυτή. Εκφράζουμε ιδιαίτερε ανησυχίες όμως τώρα όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των δύο εταιριών γιατί ακριβώς μετά το Φεβρουαρίου η Gazprom αποφάσισε να σταματήσει τις συμβάσεις εφοδιασμού και την μεταφορά του φυσικού αερίου. Αν όντως σταματήσει ο εφοδιασμός αυτός, θα έπρεπε να γίνει συντεταγμένα, λαμβάνοντα υπόψη τι υποχρεώσει και των δύο πλευρών και τα δικαιώματα και των δύο πλευρών, αλλά και τι επιπτώσει σε τρίτε χώρε, όπω για παράδειγμα στι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι είναι προ το συμφέρον όλων και η Gazprom και η Ναυτογκάς και η Ρωσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθήσουν την απόφαση τη διαιτησία τη Στακχόλμη. Δεν πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση από καμία πλευρά. Και είναι ακόμα δυνατόν η Γκάσπρομ να συμμορφωθεί με την απόφαση και να πληρώσει τα 2,6 δισεκατομμύρια ε, αμερικανικά δολάρια στην Ναυτογκάς και να προβεί στον εφοδιασμό φυσικού αερίου. Και ε, περιμένουμε από τις Ουκρανικές Αρχές και την Αυτογκάς να δράσουν υπεύθυνα και να συνεχίσουν να μεταφέρουν το φυσικό αέριο παρά τις δυσκολίες. Πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει διακοπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη να διευκολύνει τις συνομιλίε στην τρέχουσα κατάσταση. Όπως ξέρετε, η Ουκρανία την 1η Μαρτίου ξεκίνησε τον μηχανισμό έγκαιρη προειδοποίησης βάσει τη Συμφωνία Σύνδεση όταν έπαψε να εφοδιάζει, να εφοδιάζει την αυτογκάς. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε αμέσω και είχαμε διμερεί διαβουλεύσει με τον Πρωθυπουργό τη Ουκρανία, τον κύριο Γκρόισμαν, με τον ε, Διευθύνοντα Σύμβουλο τη Ναύτογκα, τον κύριο Κομπόλεγεφ και τον Υπουργό Ενέργεια τη Ρωσία, τον κύριο Νόβακ. Επίσης υπήρξαν και τεχνικέ διαβουλεύσεις μεταξύ των διαφόρων πλευρών. Συνεχίζεται ο διάλογο πάντως και με την NSOG προκειμένου ελέγξουμε πώς προχωράει η κατάσταση. Όσον αφορά τώρα την σύμβαση μεταφοράς που, εκπνέει μάλλον το 2019, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τριμερείς συνομιλίες όσο γίνεται πιο γρήγορα προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για το τι θα γίνει με την μεταφορά όγκων μετά το 2019. Η αποσύνδεση και ο εξυγχρονισμός του δικτύου μεταφοράς είναι βασικά στοιχεία. Και θα συνεργαστούμε και με τις Ουκρανικές Αρχές και την Αύτογκας για να προχωρήσουμε στην αποσύνδεση. Η ανάμιξη ε, επιχειρήσεων δυτικών στις οποίες έχουμε εμπιστοσύνη μπορεί να βοηθήσει στην ασφάλεια όλων μας μετά το 2019 για την μεταφορά αυτή. Όλες οι πλευρές έχουν να κερδίσουν από αυτό. Η ασφάλεια ενέργεια στην Ευρώπη εξαρτάται πολύ από την καλή λειτουργία, από τη διαφάνεια, στην ε, αγορά υγροποιημένης ενέργειας. Το ρυθμιστικό μας πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης και της οδηγίας για το φυσικό αέριο, προχωράει προκειμένου να προσφέρει ισορροπά και να αποφεύγονται οι καταχρήσεις. Η Επιτροπή σας ε, ψήφισε σχετικά τροπολογία σήμερα το πρωί. χώρο της τροποποίησης που πρότεινε τον περασμένο Νοέμβρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να διευκρινίσει την, το ότι η νομοθεσία μας ισχύει για όλες τις, όλους τους αγωγούς και όλες τις γραμμές διασύνδεσης μέχρι τα όρια ελέγχου της Ένωσης. Έτσι θα διασφαλίσουμε ότι όλοι οι αγωγοί εισάγονται που μπαίνουν στην Ένωση συμφωνούν με τους κανόνες μας και λειτουργούν με διαφάνεια και είναι διαθέσιμοι και για άλλους επιχειρήσεις και λειτουργούν αποτελεσματικά. Όπως είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ στην επιστολή προθέσεων που ε, συνόδευε την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης είναι σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ένωσης και θα ενισχύσει ιδιαίτερα την ε, διάσταση αλληλεγγύης, δημιουργώντας ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μεταφορά της Ένωσης στην Ένωση ανεξαρτήτως προέλευσης. Οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θετική σας ψήφο, την υπερψήφιση της τροποποίησης και ελπίζω το Συμβούλιο να ολοκληρώσει τη θέση του με βάση την πρότασή μα, ώστε ο τριμερής διάλογο να αρχίσει να τον πιο σύντομα. Θέτω το θέμα αυτό σε κάθε επίπεδο και σε επίπεδο πρωθυπουργών ε, και σε επίπεδο του Υπουργού Ενέργειας της Βουλγαρίας στην τελευταία μου επίσκεψη στη Σόφια όταν συζητούσαμε το θεματολόγιο της Βουλγαρικής Προεδρίας και ξέρω ότι ο κύριος Πρόεδρος επίσης θα πάει στη Βουλγαρία πολύ σύντομα ελπίζουμε λοιπόν όλοι ότι οι εκκλήσεις που κάνουμε προς την Προεδρία, ιδιαίτερα μετά από την ευρεία στήριξη που πήρε η τροπολόγηση αυτή στην Επιτροπή σας, θα οδηγήσει σε ταχεία κατάληξη του θέματος αυτού στο Συμβούλιο και σε έναρξη της τρεμερούς διαδικασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμποδιομητική σας στάση έναντι της προτάσεως αυτής για τροποποίηση και ελπίζω ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον για να καταλήξουμε σε ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. για τις παρατηρήσεις που κάνετε για τα θέματα αυτά, για την παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Πολύ σημαντικό θέμα για μας όπως είπατε. Είμαστε πολύ κοντά στην Ουκρανία. Και είμαστε στενά συνδεδεμένοι σε πολλούς τομείς με την Ουκρανία. Είμαστε εταίροι. Είναι πολύ σημαντικός εταίρος. Γιατί πρέπει όλοι να δρουν με υπεύθυνο τρόπο. Στις διεθνείς σχέσεις χρειαζόμαστε υπευθυνότητα. Αλλιώς όλα θα καταρρεύσουν. Λοιπόν, να αρχίσουμε τη συζήτηση. Πρώτα από το ΕΛΚ. Ο συντονιστής Χριστιανής Κάρης. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωστή η δέσμευσή σας για τα θέματα αυτά. Και χαίρομαι που ήρθατε και πάλι στην Επιτροπή μας, αλλά ε, είναι ατυχής η στιγμή για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Θα αρχίσω με το σχόλιο και μετά θα κάνω ερώτηση. Το σχόλιο. Το, το ότι είναι ατυχής η συγκυρία δεν είναι και τόσο σπάνιο. Η ρωσική κυβέρνηση και στο παρελθόν, επειδή έχει αυτό το κρατικό μονοπόλιο την Gazprom, αξιοποιεί ως πολιτικό όπλο την παροχή αερίου. Μετά την ε, απόφαση της διαιτησίας στη Στοχόλμη που σήμαινε ότι θα έπρεπε να πληρώσει η Gazprom ε, πολλά λεφτά στην Αυτογκάζ, αντί να αρχίσουν να πληρώσουν, αντί να πούνε να ένα χρονοδιάγραμμα για τις ε, πληρωμές, κόψανε την παροχή αερίου στην Ουκρανική αγορά. Τη στιγμή που υπήρχε τρομερό ψύχος, παγετός. Οι Ουκρανοί χρειάστηκε να κλείσουν τα σχολεία τους για να διασφαλίσουν την ε, παροχή φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά αυτό είναι εντελώς αντίθετο από ότι στο κράτος δικαίου. Το, η διατησία λέει πληρώστε και εσύ το αντίθετο. Γιατί ξέρετε, ότι η στάση της ρωσικής κυβέρνησης ότι χρησιμοποιεί, αξιοποιεί την κάθε ως πολιτικό όπλο αξιοποιείται κατά των πιο αδυνάμων φυσικά, του πιο αδύναμου κρίκου. Δεν είναι μέλος της Ένωσης η Ουκρανία, μπορεί να παίξει το ζόρικο η Ρωσία και το κάνει. Με την Ευρώπη είναι πιο δύσκολο γιατί παίρνει πολλά λεφτά για το αέριο από την Ευρώπη. Όπως σωστά είπατε, η Επιτροπή μας με ιδιαίτερα ευρία πλειοψηφία στήριξε την προώθηση της βελτίωσης που πρότεινε η Επιτροπή για την οδηγία για το αέριο. Και φυσικά, αν περάσουν οι προτάσεις μας στο, τριμερές, ε, στο τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο, θα αυξηθεί η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμμετάσχει ενεργά σε προγράμματα και εγχειρήματα που θα διασφαλίσουν τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων και που θα επιτρέψουν ουσιώδη άσκηση ενεργειακής πολιτικής. Ερωτήσεις. Πώς θα αντιμετωπιστεί μέσω του τρομερούς διαλόγου από το Συμβούλιο αυτή η οδηγία και δεύτερον, πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δικαιολογημένες ανησυχίες των συναδέλφων από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία που ανησυχούν πολύ ότι η οδηγία αυτή θα αποτελέσει εμπόδιο στην κατασκευή αγωγών από τη Βόρεια Αφρική και αν, ε, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν προβλήματα για παράδειγμα με τη Λιβύη αν θες να συζητήσεις την κατάσταση με τη Λιβύη δεν ξέρεις ούτε καν με ποιον να μιλήσεις γιατί δεν ξέρεις ποιος ε, διοικεί τη χώρα γίνονται μάχες δεν είναι σαφές ποιος διοικεί, ποιος επικρατεί είναι δικαιολογημένες αυτές οι ανησυχίες των ε, Νοτιοευρωπαίων. Τι θα γίνει με τα υπάρχοντα συμβόλαια, ενισχύ συμβόλαια. Εάν εγκριθεί αυτή η οδηγία και γίνει νόμο, πώ θα επηρεάσει, εάν επηρεάσει, τα ισχύοντα, τις ισχύουσες συμβάσει για παρχαίριο. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενο ομιλητή από του σοσιαλιστέ ε, ο συντονιστής Νίκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Σεύκοβιτς για την ε, παρουσία του και να τον ευχαριστήσω για τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ύψης της σημασίας το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Και αυτό το εκτιμούμε ιδιαίτερα ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπου δυστυχώς βλέπουμε ότι η πρόσβαση σε φυσικό αέριο ε, ε, βασίζεται σε ένα παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων, μιας μεγάλης δύναμης, τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ε, συνθήκες ψύχους που πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον πληθυσμό. Θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την οδηγία περί φυσικού αερίου. Ποιος θέλει να συνάψει συμβα... Όποιος θέλει να συνάψει συμβάσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τηρεί όλες τις ε, προδιαγραφές. Αυτό είναι απόλυτα σαφές και νομίζω ότι όλοι ακούσαμε αυτό το μήνυμα, το οποίο είναι ένα στεναρό μήνυμα προς τη Ρωσία. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι πριν από δύο εβδομάδες δεν έγινε ε, κατανοητό το θέμα της ενεργειακής ενέργειας με βάση τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί μιλάμε για μια στοχοθέτηση η οποία ετέθηκε από το Συμβούλιο του 30% και δυστυχώς αυτό δεν έγινε κατανοητό από πολλά κράτη-μέλη. Και αυτό το μήνυμα ήταν στεναρό. Τώρα, σε σχέση με τη Ρωσία και την Ουκρανία, αυτή την ε, περίπλοκη θέση, η θέση της Επιτροπής είναι πολύ σωστή, αλλά θα πρέπει να έχει και συνέχεια, γιατί φυσικά έγινε αυτή η διαιτησία, η οποία όμως ε, φαίνεται ότι δεν τηρείται. Δηλαδή, μερικοί θέλουν ειδικέ σχέσεις και ειδική μεταχείριση, παρά τις αποφάσεις ενός διεθνούς δικαστηρίου διατησίας. Τώρα, σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να προσδώσουμε σημασία στις περιφέρειες που βασίζονται στο φυσικό αέριο. Και εδώ θα μιλήσω για τη Μαύρη Θάλασσα. Εδώ υπάρχουν και κοιτάσματα φυσικού αερίου πολύ υψηλότερα από τις ανάγκες της Ρουμανίας. Θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες και της ε, Ουγγαρίας και της Αυστρίας καθώς και της ε, Τσεχίας. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει διαφοροποίηση αυτής της στρατηγικής ως προς τον εφοδιασμό. Θα εργαζόμαστε με μεγάλη ευθύνη σε αυτό το θέμα και ως προς τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ελαφρά την καρδία. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για την ε, δική σας προσωπική ανάμειξη. Ευχαριστώ. Και βεβαίως θα μπορούσατε να εφοδιάσετε και τη ε, Βουλγαρία πέρα από την ε, Ουγγαρία και την ε, Αυστρία, καθώς και την Τσεχία που είπατε. Ο κύριος Στοσανόφσκι. Έχετε το λόγο από πλευράς συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ευχαριστώ πολύ και εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο Επίτροπος μας επισκέφθηκε ε, μετά το 2006 και το 2009 Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο και έκτοτε έχουμε βρει σοβαρές τεχνολογικές λύσεις, μετά το 2006 δηλαδή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρκετά ασφαλής. Δεν έχουμε πληγεί ιδιαίτερα. Βεβαίως αυτή τη φορά δεν θα ακούσετε απλές ερωτήσεις και ίσως και οι απαντήσεις σας να είναι δύσκολες γιατί θα σας μιλήσουμε και για τρίτες χώρες. Χαίρομαι γιατί προχωρήσαμε πολύ μετά το 2006 με την αντίστροφη αυτή ροή ως προς την Τσεχία και τη Σλοβακία. Τώρα υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού. Γιατί μιλώ για θέματα δύσκολα. Όταν ε, ολοκληρωθεί και το North Stream 2, η κατάσταση για την Ουκρανία θα είναι ακόμα πιο δυσχερής υπό την έννοια των συμβατικών σχέσεων, γιατί το North Stream 2 θα προβάλλει πολλές αλλαγές και θα υπάρχει άλλη διέλευση. Δεν θα χρειάζεται πια η διαμετακόμιση, η διέλευση αυτή όπως την χρειαζόμασταν μέχρι τώρα. Και γι' αυτό θα πρέπει ίσως να αποζητήσει νέες τεχνολογικές λύσεις. Μετά το North Stream 2 η κατάσταση θα είναι εντελώς διαφορετική. Τώρα έχουμε ακόμα ε, χρόνο για σκέψη ως προς τα δίκτυα διασύνδεσης, αλλά μετά το North Stream 2 η κατάσταση θα είναι εντελώς διαφορετική. Τώρα, ως προς τις τρέχουσες συζητήσεις για το ενεργειακό πακέτο, η μεγαλύτερη εξάρτηση από τρίτες χώρες ως προς το φυσικό αέριο, όπως το είχαμε ζήσει με τον άνθρακα και άλλα ορυκτά καύσιμα στο παρελθόν, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο λοιπόν θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για το μέλλον βασιζόμενοι στο παρελθόν. Είναι πολύ δύσκολες οι ερωτήσεις, είναι πολύ εύκολο να τις θέτει κανείς, αλλά δύσκολο να βρεθούν οι σωστές απαντήσεις. Ευχαριστούμε πολύ για την ερώτηση. Ο επόμενος ομιλητής εξ ονόματος των Πρασίνων, ο Κλοντ Τούρμες, ο συντονιστής. Ευχαριστώ κύριε Μπούζεκ. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Βρισκόμαστε σε μία φοβερή κατάσταση ένας ε, ουκρανικός φορέας, η επιχείρηση που έχει προπληρωθεί, έτσι ώστε σε καταστάσεις ψύχους να μην πληγεί ο πληθυσμός, βλέπουμε ότι ο αντίστοιχος ρωσικός φορέας 15 λεπτά μετά από τον εφοδιασμό αποφασίζει να μην προμηθεύσει εκθέτοντας ε, γυναίκες, παιδιά και ανθρώπους μεγάλης ηλικίας ε, να είναι εκτεθειμένοι στο ψύχος. Και ο ίδιος, η ίδια επιχείρηση, ο ίδιος φορέας μείωσε την πίεση παροχής αερίου έτσι ώστε να υπάρχει ενός τύπου εσωτερική έκρηξη του ουκρανικού φυσικού αερίου. Αυτό έγινε σκόπιμα για να ε, μην μπορεί να λειτουργήσει το δίκτυο της Ουκρανίας σε περίπτωση μη παράδοσης και μη εφοδιασμού. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μια στεναρή απάντηση. Έχω λοιπόν μια συγκεκριμένη ερώτηση προς εσάς ε, σε σχέση με αυτή τη συμφωνία ε, διέλευσης ε, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που λύγει το 2021 νομίζω αφορά θέματα της ε, Επιτροπής αλλά και της Γαλλίας και της Γερμανίας γιατί με βάση τη Συμφωνία του Μίνσκ θα πρέπει να υπάρξει και μία μεταγενέστερη συμφωνία με τη Ρωσία. Σήμερα δεν μου κάνει εντύπωση που οι κομμουνιστές αυτού του οίκου βρίσκονται στο μέρος της ε, Ρωσίας και οι ακροδεξιοί πληρώνονται από τον Πούτιν. Αλλά είμαι περήφανος γιατί εμείς οι πράσινοι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες έχουμε σαφή θέση. Αυτό αφορά και τους ε, Πολωνούς που είναι με το Γέρσι Μπούσεκ αλλά και η πράσινη της Γερμανίας Ρεμπέκα είναι η μόνη που μας υποστηρίζουν και οι πράσινοι στη Γαλλία, κυρία Γκροστέτ, έχουν μία σαφέστατη θέση. Και αν έχω να αποστείλω ένα μήνυμα στη γαλλική κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε Μακρόν, είναι απαράδεκτο μία γαλλική κυβέρνηση που υπέγραψε τη συμφωνία του Μίνσκ ε, στην ουσία υποσκάπτει την οικονομική υγεία και στεναρότητα της Ουκρανίας σε αυτό το θέμα. Ελπίζω να ε, ε, γίνει αυτό δεκτό. Ο κύριος Μάστρελικ ήταν αυτός ε, ο οποίος επέβαλε κάτι τέτοιο στον κύριο Ολάντ. Ελπίζω ο κύριος Μακρόν να μην υποσκάπτει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε αυτό το θέμα. Thank you very much, uh, Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, εκ μέρους της ΓΚΟΕ, ο κύριος Μπενίτου Ζιλουάγκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τον Επίτροπο Σεύκοβιτς που ήρθε σήμερα στην Επιτροπή μας. Θέλω να εκφράσω μία ανησυχία μου, η οποία δεν ξέρω αν έχει να κάνει μόνο με την κοινωνία στην Ουκρανία, έχει να κάνει και με τον κίνδυνο που ελοχεύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά που μας είπατε και ανησυχία σας έχει να κάνει με την ασφάλεια εφοδιασμού. Το θέμα της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο θέτεται, αλλά όχι την εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο γενικά, είτε πρόκειται για ρωσικό είτε για οτιδήποτε άλλο. Για να αποφύγουμε αυτή την εξάρτηση, είπατε ότι χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια στις συμφωνίες, στις συμβάσεις των χωρών μελών, τη διαφοροποίηση των πηγών, το κοινό συμφέρον στη διαφοροποίηση κτλ. Αλλά έχετε θέσει ποτέ υπομφισβήτηση το ίδιο το φυσικό αέριο και την σχέση του με την κλιματική αλλαγή. Λαμβάνετε υπόψη σας εκπομπές μεθανίου. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσο σκέφτεστε να αναθορίσετε και τους ε, στόχους άλλων ενεργειακών μέτρων, όπως είναι η οδηγία για τις ανανεώσιμες, ε, την ενεργειακή επάρκεια. Μήπως σκέφτεστε να αναθεωρήσετε και αυτούς τους στόχους, έτσι ώστε να συνάδουν με τη στρατηγική αυτή μείωση εξάρτησης, όχι μόνο από το ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά από το φυσικό αέριο γενικώ. Υπήρξε ένα non-paper από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μιλούσε για την ε, αναθεώρηση ώστε να χρησιμοποιούνται περισσότερο νόσιμες ενέργειες. Γίνεται αυτό και στα πλαίσια της ενεργειακής επάρκειας. Θα βοηθούσε πολύ την καταπολέμηση της εξάρτησής μας αυτής από το φυσικό αέριο και της Ρωσίας. Έπειτα υπάρχουν διάφορες μεγάλες ε, επιχειρήσεις, ευρωπαϊκές, η ταλ ας πούμε, η γαλλική που έχει το 20% ε, στη Βόρεια Ρωσία για το υγροποιημένο φυσικό αέριο ε, και άλλοι που συμμετέχει στο North Stream 2 για παράδειγμα. Στις συναντήσεις με τις επιχειρήσεις αυτές, για τι πράγμα μιλάτε τελικά. Πώς εξηγείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρά τις στενές σχέσεις που έχει με αυτές, δεν μπορεί να επιβραδύνει την ε, διαδικασία για τον νέο αυτό ρωσικό αγωγό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Χάρμς. Es gab ja in den letzten Tagen, there were during the last days äh, also. Τις τελευταίες ε, μέρες Είδαμε και διάφορα για διμερείς συναντήσεις Ουκρανίας-Ρωσίας για τα προβλήματα που προέκυψαν από τότε που μείωσε την πίεση στον αγωγό η Ρωσία. Ξεκίνησε δηλαδή επίσημα ε, μια τριμερής ε, σχέση εξαιτία της ε, κρίσης αυτής. Όντως είναι μια εκτακτή κατάσταση και γι' αυτό πρέπει να έχουμε τριμερείς συναντήσεις όπου να συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί να προτείνει καλύτερες λύσεις από τις διμερείς. Θέλω να ξέρω λοιπόν ποια είναι η δικιά σας θέση από αυτού. Και θα ήθελα να ακούσω και κάτι για το εξή. Υπάρχει αντίδραση, προβληματισμός στη θέση του Συμβουλίου προκειμένου να ρυθμίσει την αγορά φυσικού αερίου, έτσι όπως αρχίσαμε σήμερα να συζητάμε στην Επιτροπή μας. Υπάρχει τέτοια σκέψη μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με την Ουκρανία. Ή συνεχίζουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και οι Γερμανοί και οι άλλοι παίζουν τα δικά τους στα χαρτιά όπως έχουν κάνει και κατά το παρελθόν. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω στον συνάδελφο Τουρμές ότι έχω βαρεθεί αυτά τα μαθήματα ηθικής. Πολλά θα μπορούσα να πω για το Λουξεμβούργο, αλλά δεν το κάνω ποτέ. Οπότε να προσέχει τι λέει. Στη συνέχεια, για το θέμα που μας αφορά, θέλω να επενθυμίσω ότι πάντα ήθελα να στηρίξουμε τον διπλό στόχο που είναι η ασφάλεια εφοδιασμού και από την άλλη διαφοροποίηση των πόρων. Σας άκουσα κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, μας είπατε ότι το φυσικό αέριο είναι βασικό σε αυτή τη μεταβατική περίοδο όπου οι ανανεώσιμες ενέργειες δεν μπορούν να διασφαλίσουν τον αναγκαίο εφοδιασμό. Εξάλλου το λέω γιατί πράσινοι αρνούνται τα ορυκτά, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την ανάγκη ότι χρειαζόμαστε αέριο. Τι γίνεται τώρα με την εταιρική μας σχέση με την Αφρική, γιατί συστηματικά μιλάμε για την Gazprom, για τον εφοδιασμό φυσικού αερίου ρωσικού, αλλά η διαφοροποίηση τι σημαίνει. Υπάρχει φυσικό αέριο και στην Αφρική. Πού βρισκόμαστε από αυτού. Θα ήθελα να μου πείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κόχλιτσεκ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Έχω κάποια σχόλια. Δεν θα σχολιάσω τις ανοησίες που εξτόμησε ο κύριος Τούρκος αυτά πιστεύει, αυτές είναι απόψεις του και έχει κάθε δικαίωμα να τις πιστεύει. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Δεν μας ανησυχεί ότι από τη Λιβύη έχουμε ένα μόνο προμηθευτή. Είναι μονοπόλιο δηλαδή. Και δεν ξέρουμε και ποιος είναι. Και από την Αλγερία επίσης υπάρχει ένα μονοπόλιο προμηθευτής μας. Στην Αλγερία είναι προφανές ότι μόνο μονοπωλιακή μπορεί να είναι μονοπωλιακός ο εφοδιασμός μας. Και δεν μας πειράζει. Γιατί η Ρωσία μας πειράζει. Και επιπλέον, γιατί η Κομισιόν δεν ασχολείται με το φυσικό αέριο που μπορεί να εξαχθεί από τις θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Κύπρο. Γιατί μας υποβάλλουν αυτές τις ερωτήσεις. Ξέρω ότι είναι περίπλοκη η κατάσταση γιατί Υπάρχει το πρόβλημα της Τουρκίας και της Βόρειας Κύπρου, αλλά παρόλα αυτά. Τρίτη ερώτηση. Ποιος από την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν κατά της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου για τους φτωχούς στην Ουκρανία. Τρεις φορές. Δεν άκουσα καμία διαμαρτυρία κατά αυτού. Από κανέναν. Ούτε από του πράσινου, ούτε από το Κοινοβούλιο, την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και κάτι ακόμη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Όταν, για παράδειγμα, ήρθαν οι κυρώσεις κατά του Ιράν, γιατί το Ιράν είναι από τους κυριότερους προμηθευτές φυσικού αερίου. Και υπάρχει ο αγωγό μέσω Τουρκία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αγοράσουμε φυσικό αέριο από το Ιράν, αλλά δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό. Και τελευταίο, οι πράσινοι αδελφοί μα πραγματικά πιστεύουν ότι το μεθάνιο είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Γιατί είναι και αεροθερμοκηπίου, ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε πρόεδρο. Ο κύριο Μπούτιχόφερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε την Πρόεδρε, για την πληροφόρηση αυτή. Εγώ διαφωνώ με την κυρία Γκροστέτ, γιατί με εξέπληξε όταν αντέδρασε σε μια πολιτική επίκριση. Διότι αντέδρασε στις επικρίσεις του κυρίου Τούρμες με εθνικιστικά σχόλια. Του επιτεθήκατε επειδή είναι Λουξεμβούργιος. Δεν σε επιτέθηκε σε εσά επειδή είστε Γαλλίδα. Επέκρινε την πολιτική της Γαλλίας, γιατί είναι λανθασμένη είναι λαθασμένη και από ενεργειακής και από γεωπολιτικής και από περιβαλλοντικής πλευράς. Δεν είναι σωστό στο κοινοβούλιο μας εάν κάποιος επικρίνει τη γαλλική πολιτική, μία γαλλική πολιτική, να αντιμετωπίζεται με τέτοιες ε, εθνικιστικές ε, κορώνες. Θα παρακαλούσα τη Γαλλική Δημοκρατία Μπορείς να, μπορείτε να φύγετε αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, αλλά θα το πω. Αλλά έχω κάθε λόγο να το πω. Και επικρίνω πολύ συχνά και τη δική μου κυβέρνηση. Τώρα όμως επικρίνω τη δική σας. Ο πρόεδρος, παρακαλώ, ηρεμήστε. Είναι θέματα ασφάλεια τη Ευρώπη τα θέματα αυτά. Δεν το καταλαβαίνει η γαλλική κυβέρνηση. Είναι θέματα συνοχή τη Ευρώπη. Είναι θέματα διαμόρφωση του μέλλοντο τη Ευρώπη από του ίδιου του Ευρωπαίου. Όσο δεν το καταλαβαίνει αυτό το Παρίσι και άλλες κυβερνήσεις δεν έχει καμία έννοια η ευρωπαϊκή ενοποίηση γιατί με το θέμα αυτό προκαλούμε διχασμούς μεταξύ ανατολικών και δυτικών χωρών. Προκαλούμε διχόνοια στην Ευρώπη. Γιατί πάντα διακηρύσουμε ότι η Ευρώπη σημαίνει αλληλεγγύη, αλλά όταν τα ανατολικά κράτη-μέλη του αλληλεγγύη, ξαφνικά δεν γίνεται τίποτα. Ο πρόεδρος, παρακαλώ ηρεμήστε να συζητάμε με επιχειρήματα. Θέλει κανείς άλλο τον λόγο. Δεν ξέρω μήπως η κυρία πρώτη, επειδή είναι η κυρία... Α, θέλει η Ρεμπέκα. Ας δώσουμε χρόνο στον ε, αντιπρόεδρο να απαντήσει, γιατί ε, ε, έχει ε, πολλές ερωτήσεις να αντιμετωπίσει. Θα ήθελα να ζητήσω από τους πρασίνους συναδέλφους το εξής. Βεβαίως, όλοι έχουμε συναισθήματα, αλλά η κυρία Γκροστέτ ε, δεν ε, ακολουθούσε αυτό το, το δρόμο που εσείς είπατε. και δεν λοξοδρόμησε. Όταν έχουμε συναισθήματα δεν είναι σκόπιμο να τα μεταφέρουμε ή να επιθέμεθα ο ένας τον άλλον. Έχουμε τον Επίτροπο ενώπιόν μας, άρα δεν έχει νόημα να εκφράζουμε τις προσωπικές μας απόψεις. Ίσως θα πρέπει λοιπόν να επιβραδύνουμε αυτούς τους ρυθμούς και αυτές τις αντιδράσεις. Ο Αντιπρόεδρος έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω τα ερωτήματα των Ευρωβουλευτών, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να διασαφηνίσουμε τα θέματα που προέβαλαν. Ο κύριος Κάρινς ρώτησε πώς θα περάσει το ζήτημα στο Συμβούλιο, πώς θα αντιμετωπιστεί με βάση τις πρόσφατες συζητήσεις με τη Βουλγαρική Προεδρία. Ε, τους εξήγησα ακριβώς ότι θα πρέπει να ε, παραμερίσουμε νομικίστικες ε, προσεγγίσεις. Έχουμε τις νομικές υπηρεσίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου που κονταροχτυπιούνται και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία νομική βάση με βάση την ε, εδαφική της έκταση. Άρα ξέρουμε πού και πότε πρέπει να εφαρμοστεί ένα νομικό πλαίσιο και έκανα μια έκκληση προς τη Βουλγαρική Προεδρία να αποτελέσει εμπροστοφυλακή. Θα πρέπει να επιλύσουμε αυτή την νομική διαμάχη και να φτάσουμε σε ένα έγγραφο, αναθεωρημένο έγγραφο υπαριθμών 1, που θα μπορέσει να προετοιμάσει η Γραμματεία του Συμβουλίου και θα συζητηθεί από τα κράτη-μέλη. Πολλά κράτη-μέλη θα ήθελαν να το συζητήσουν και η συζήτηση θα μπορούσε να ακολουθήσει δύο γύρους. Στο πρώτο μέρος θα προετοιμαστεί η εργασία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και στόχος μας είναι να φτάσουμε σε μια γενική προσέγγιση στο τέλος της Βουλγαρικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Υπουργών Ενεργείας του Ιουνίου. Χάρηκα λοιπόν για τη σημερινή σας ψήφο, γιατί ε, φαίνεται ότι το ένα νομοθετικό σκέλος συνδράμει το άλλο. Έτσι ώστε και το Συμβούλιο να ξεκινήσει μια συζήτηση πέραν από τις συμβουλές της νομικής ε, υπηρεσίας, γιατί φυσικά έχει μεγάλη σημασία η νομική υπηρεσία, αλλά έχει συμβουλευτικό ρόλο. Θέλουμε μια συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο και μια επικοδομητική προσέγγιση έτσι ώστε στον τριμερή να δώσουμε τελική μορφή σε αυτή την τροποποίηση η οποία δεν είναι και τόσο ε, δυσχερής. Θέλουμε να δούμε πώς η οδηγία περί φυσικού αερίου θα εφαρμοστεί, γιατί υπάρχουν πολλές αποκλήσεις από τη νομική υπηρεσία και γι' αυτό, ε, αυτό ακριβώς υπήρξε τροχοπέδι στις εργασίες μας. Θα συνεργαστούμε με τη Βουλγαρική Προεδρία με βάση το έγγραφο αυτό την πρώτη αναθεώρηση έτσι ώστε να δώσουμε μια όθηση στις συζητήσεις ως προς τις συγκεκριμένες ερωτήσεις των Ιταλών, των Ισπανών και άλλων συναδέλφων θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν σαφείς απαντήσεις προς όλους και προσπαθούμε να ε, δίνουμε άμεσες απαντήσεις και διμερώς με τις χώρες, γιατί πάντα υπάρχουν καλές λύσεις για όλους ε, τους αγωγούς. Μπορούμε να δουλέψουμε με εξαιρέσει, να λάβουμε υπόψη την κατάσταση στη Λιβύη. Δεν ξέρουμε με ποιον συνομιλούμε εκεί. Και θα ήθελα να γίνουν διαβουλεύσεις με όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θέλουν διασαφηνίσεις γιατί όλα τα προβλήματα μπορούν να επιληθούν. Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε διοικητικά την κατάσταση. Θα πρέπει όμως να έχουμε ενιαία εφαρμογή του νομικού πλαισίου περιφυσικού αερίου. Κύριε Νίκα, σας ευχαριστώ πολύ για τα ευγενικά σας σχόλια και την αξιολόγησή σας ως προς την ενεργειακή ασφάλεια. Χτες βρέθηκα στην Διατλαντική Συμμαχία, στη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ και είδα ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι ε, τρία χρόνια πριν εξαιτίας των ε, δοκιμών αντοχής επειδή έχουμε κάνει επενδύσεις υποδομών και αντιστρόφων ρών και επειδή ακριβώς δώσαμε ε, όθηση σε θέματα και ε, ε, υποδομών και λογισμικού για να μην γνωρίσουμε την κατάσταση του 6 ή του 9. Γι' αυτό σας ευχαριστώ πολύ για αυτά τα προγράμματα κοινού ενδιαφέροντος. Ε, διαφορετικά θα είχαμε τη συνέχεια μιας ε, κατακαιρματισμένης αγοράς όπου δεν θα είχαμε ελεύθερη ροή ενέργειας. Αρχίσαμε με το φυσικό αέριο γιατί εκεί η αγορά ήταν πολύ κατακαιρματισμένη και ήταν υπέρ εκείνου που υπερήχε στην αγορά, που κατήχε δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα του, του ηλεκτρισμού και στο PCI που έχει σχέση και με το ενεργειακό μείγμα στην Ευρώπη. Ως προς τη Μαύρη Θάλασσα και αυτή την προοπτική που διανοίξατε, Υπάρχουν πολλά διερευνητικά προγράμματα από τη Ρουμανία αλλά και τη Βουλγαρία και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο αυτές οι δύο ε, χώρες αλλά τα Δυτικά Βαλκάνια, η Μολδαβία και οι πρώην ανατολικές χώρες να μπορέσουν να προβούν σε αυτή την αποτίμηση που άρχισε πριν από τρία χρόνια. Γιατί θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα κοιτάσματα στη Μαύρη Θάλασσα, έτσι ώστε να διανοίξουμε και αυτές τις αγορές. Δεν πρέπει μόνο να ε, γίνει αυτή η σύνδεση Βουλγαρίας-Ρουμανίας γιατί έχει ήδη γίνει αυτή η διασύνδεση αλλά να χρησιμοποιηθεί σωστά. Η Βουλγαρία με τη δική μας βοήθεια θα πρέπει να βελτιώσει την ποιότητα των εσωτερικών αγωγών στο δικό της έδαφος γιατί έτσι θα μπορέσει να προβεί όχι σε διαμετακόμιση, αλλά να είναι εμπορικός και οικονομικός φορέας, ο οποίος θα παράσχει καλές υπηρεσίες σε όλες τις γειτονικές χώρες. Αυτό ακριβώς είπα στη Σόφια και αυτό αφορά τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Να υπάρχει αυτή η συνδεσιμότητα η οποία εκλείπει. Εάν συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, θα επιβεβαιώσουμε ότι κάθε χώρα θα έχει πρόσβαση σε τρεις πηγές φυσικού αερίου και δεν θα υπάρχει δεσπόζουσα θέση. Και αυτό είναι καλύτερο για την διαπραγμάτευση τιμών, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και θέλω να το τονίσω για άλλη μια φορά. Όπως είπατε και εσείς, πολλά χρόνια, για πολλά χρόνια, και νομίζω και τα στατιστικά στοιχεία του 2015 δείχνουν ότι η τιμολόγηση για τις ανατολικές χώρες είναι πολύ ψηλότερη από ότι για τις δυτικές, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται πολύ ε, πιο κοντά στην πηγή φυσικού αερίου. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνδεσιμότητα για να είμαστε δίκαιοι προς όλα τα μέλη τα οποία θα μπορέσουν να καρποθούν από την ενεργειακή πολιτική της εσωτερικής αγοράς. Κύριε Τοσενόφσκι, θα σας απαντήσω σλοβακικά, αν μου επιτρέψετε. Και το ίδιο κάνω και με τους τσέχους φίλους. Η συνεργασία με την Ουκρανία έχει μεγάλη σημασία γιατί έχουμε αποτιμήσει την κατάσταση και με βάση την τελευταία κρίση φυσικού αερίου του 2009 είδαμε ότι η Σλοβακία σώθηκε επειδή ακριβώς υπήρξε αντίστροφη ροή αυτή ήταν δηλαδή η λύση που δόθηκε από, τους, ε, από τα ευρωπαϊκά κομβικά σημεία. Και είχαμε αυτή την εμπειρία και για την ε, Ουκρανία. Γιατί υπάρχει δυνατότητα αντίστροφης ροής και από την Πολωνία και ε, από την Ουγγαρία. Η Ουκρανία δεν αναγκάστηκε να αγοράσει άμεσα φυσικό αέριο από την Gazprom. Μπορεί να το αγοράσει με καλύτερη τιμολόγηση μέσω ημών. Και αυτό ακριβώς έχει μεγάλη σημασία αυτή η αντίστροφη ροή που βλέπουμε στους αγωγούς διασύνδεσης. Αυτό που έχει σημασία για το μέλλον επίσης είναι το εξής. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έργα υποδομών και στα έργα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτούς τους παράγοντες. Γιατί αυτά είναι τα στρατηγικά σημεία και αν ε, δούμε το φυσικό αέριο όπως ε, και τα ορυκτά καύσιμα βλέπουμε ότι το φυσικό αέριο, όπως είπε και ο εκπρόσωπος των Πρασίνων, δεν ε, έχει τόση μεγάλη, δεν προσφεύγει σε τόσο υψηλή χρήση του ανθρώπου άνθρακα όπως τα ορυκτά καύσιμα αφορά μία ποσοστιαία αναλογία 50% χαμηλότερη. Γι' αυτό υπάρχει και όλο ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το φυσικό αέριο. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν θέλουν καν να χρησιμοποιούν τον άνθρακα λαμβάνοντας υπόψη και τις περιβαλλοντικές πτυχές και το περιεχόμενο σε άνθρακα. Από αυτή την άποψη λοιπόν και από την πλευρά της ε, λειτουργίας του φυσικού αερίου θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει συμπλήρωμα στις ανανεώσιμες πηγές. Έτσι έχουμε μια πολύ καλή, έχουμε πολύ καλές ευκαιρίες για μακρά χρονική χρονική περίοδο. Μίλησατε και για την κατάσταση στην Ουκρανία. 30 λεπτά μετά έγινε αυτή η μεταστροφή, όπως είπε και ο κύριος Τούρμες και ο Υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας μου είπε ότι ο λόγος τελικά ήταν ότι η Gazprom δεν είχε αυτή την προσθήκη, αυτό το addendum ε, της συμβατικής υποχρέωσης κάτι το οποίο αμφισβητείται από την Αυτογκάς της Ουκρανίας γιατί είπε ότι είχε γίνει συζήτηση μεταξύ επιχειρήσεων και οι νομικές υπηρεσίες ε, αποφάνθηκαν για το πώς θα οργανωθεί και προπληρωθεί αυτή η υπηρεσία. Άρα υπάρχουν δύο εκδοχές για την κατάσταση. Από όσο ελέγξαμε, δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή να μην παραδοθεί φυσικό αέριο μέσα σε μία τόσο μικρή προθεσμία και φυσικά υπήρξε και διακύμανση της πίεσης του φυσικού αερίου στην Ουκρανία και οι Ουκρανοί τα κατάφεραν πολύ καλά να σταθεροποιήσουν την πίεση του φυσικού αερίου στους αγωγούς τους γιατί υπήρχε και αποθηκευμένο φυσικό αέριο, γι' αυτό έπρεπε να είναι πολύ δημιουργικοί έτσι ώστε να πάρουν ε, φυσικό αέριο από τις δεξαμενές και να έχουν τη σωστή πίεση στους αγωγούς. Επίσης, ε, το, στα ευρωπαϊκά σύνορα, ε, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς αερίου έπρεπε να παίξουν με αυτό το σύστημα, να είναι ταχυδακτηλουργοί κάπως και οι 48 πρώτες ώρες ήταν πολύ κρίσιμες και θα μπορούσαμε να ζήσουμε πολύ κρίσιμα σενάρια. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Είχε συμβεί πριν, αλλά τώρα ήταν πιο κρίσιμη κατάσταση. Βρισκόμασταν στο τέλος του χειμώνα, οι δεξαμενές αποθήκευσης δεν είχαν τόσο ε, πολύ φυσικό αέριο. Είχε πέσει το επίπεδο των δεξαμενών, γι' αυτό νομίζω ότι ο συνδυασμός αυτός της μικρής προθεσμίας, της βραχίας προθεσμίας, ήταν ε, κάτι το ιδιαίτερο κρίσιμο και κάτι το δυσεπίλητο, αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι συνέδραμαν και οι Ουκρανοί μείωσαν την κατανάλωση, μείωσαν τη θερμοκρασία στα σπίτια, έκλεισαν τα σχολεία, μίλησαν στη βιομηχανία που δεν κατανάλωσε. Όλα αυτά συνέδραμαν έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η πίεση. Τι θα κάνουμε για την ε, διαμετακόμιση, ως προς τη διαμετακόμιση μετά το 2020. Νομίζω ότι καθίσταται σαφές ότι μία μακροχρόνια λύση είναι να έχουν κλείσει οι προμήθειες από πολύ νωρίς για εμπορικά βιώσιμους όγκους. Θα πρέπει λοιπόν οι επενδυτές να χρησιμοποιήσουν αυτή την οδό διαμετακόμισης και να κλείνουν εκ των προτέρων αυτή την οδό διαμετακόμισης. Θα το λύσουμε τριμερός αυτό, θα το συζητήσουμε τουλάχιστον, έτσι ώστε να προασπίσουμε και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα μέσα στα πλαίσια της ε, διαμεσολάβησης. Προς τον κύριο Ζιλουάγκα θα ήθελα να πω ότι φυσικά δεν θέλουμε την εξάρτηση από το φυσικό αέριο, γι' αυτό κάναμε και προτάσεις για περισσότερες ανανεώσιμες στο ενεργειακό μείγμα για να έχουμε μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση και αυτό το είδαμε και στις συζητήσεις μεταξύ Κομισιών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και υπάρχουν πρωτοβουλίες και από το Συμβούλιο. Και με βάση τις συζητήσεις ως προς το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο Υποστηρίζουμε και το, την βασική γραμμή προώθησης του ζητήματος του ε, κλίματος ως προς το mainstreaming από δημοσιονομικής πλευράς. Για την κυρία ε, Κροστέτ, ε, φυσικό αέριο από την Αφρική. Ε, στην ουσία εισάγουμε 11% από την Αλγερία και τη Λιβύη, άρα υπάρχει, Λιβύη, άρα υπάρχει διαφοροποίηση και η Μοζαμβίκη θα ήθελε να εξάγει υγροποιημένο φυσικό αέριο και θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις εργασίες στα τερματικά και στους αγωγούς διασύνδεσης και στη Γαλλία και αυτό θα είχε μεγάλη σημασία για να έχουμε καλύτερο εφοδιασμό από αφρικανικές χώρες. Ο κύριος Κόλιτσεκ υπέβαλε ένα ερώτημα σε σχέση με την ε, Κύπρο. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν πολύ, πολλά υποσχόμενο τομέα, άκουσα ότι ίσως μπορούμε να έχουμε μια νέα Νορβηγία, εάν μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το φυσικό αέριο στη Νότιο Κύπρο. Γιατί ήδη το Ισραήλ και η Αίγυπτος ε, παράγουν μάλλον παράγεται ε, φυσικό αέριο το οποίο χρησιμοποιεί η Αίγυπτος, η Αίγυπτος και το Ισραήλ και θα μπορούσαμε να έχουμε υγροποιημένο αέριο που θα εισαχθεί στην Ευρώπη. Επίσης θα είχαμε έναν αγωγό μεταξύ Κύπρου και ε, Κρήτης μέσα στα πλαίσια ενός σχεδίου κοινού ενδιαφέροντος και μας ενδιαφέρει να δούμε ποιο θα ήταν το κόστος ε, αυτού του αγωγού για να δούμε κατά πόσο είναι βιώσιμο, αλλά θα βασιστούμε στη μεταφορά του φυσικού αερίου υπομορφή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όσον αφορά το Ιράν, επειδή είναι χώρα που χρησιμοποιεί κατά πολύ υδρογονάνθρακες, στην ουσία εισάγει πολύ μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου από το Τουρκμενιστάν έτσι ώστε ε, να μπορέσουν να αντλήσουν ε, και έχουν και μεγάλα προβλήματα με τους αγωγούς ως προς την άντληση του φυσικού αερίου. Γι' αυτό νομίζω ότι θα χρειαστούν χρόνια έτσι ώστε το Ιράν να αναπτύξει το φυσικό αέριο. Η τελευταία ερώτηση του κυρίου Μπουτικόφερ ως προς το διαχωρισμό ανατολικών κρατών και δύσης. Ελπίζω να καταδείξουμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή ενότητα όχι μόνο ως προς το North Stream 2, αλλά και στα νέα προγράμματα κατασκευής ε, αγωγών φυσικού αερίου. Νομίζω ότι έχουμε καλύτερη διαπραγματευτική δύναμη όταν μπορούμε να διαπραγματευτούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, κατακαιρματισμό της αγοράς, ιδιαίτερα μεταξύ Ανατολής Δύσης. Ελπίζουμε να χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς που έχουμε και τον ε, τετραμερή, ιδιαίτερα για την διαμετακόμιση από την Ουκρανία, έτσι ώστε να αντιπαρέλθουμε την ε, κατάσταση. Σας ευχαριστούμε. Ήταν θαυμάσια συζήτηση, ήταν εξαιρετική συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Πολύ χρήσιμη για όλους μας. Αλλά να πω κάτι άλλο. Είναι πάντα καλύτερα. Είμαι απόλυτα πεπισμένος. Πολύ καλύτερα. Να μην ε, κάνουμε προσωπικές επιθέσεις. Λόγω των ε, αποφάσεων κάποιας κυβέρνησης. Γιατί είναι τόσο σημαντικό. Θα ήθελα να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Διότι μας εκλέγουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας είμαστε υπεύθυνοι για όλες τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Έτσι έχουν τα πράγματα. Άρα δεν πρέπει και εμείς να διαφοροποιούμεθα μένα έναντι των δε και να κάνουμε προσωπικές επιθέσεις για τις αποφάσεις οποιασδήποτε κυβέρνηση. Σας παρακαλώ το έχετε υπόψη σας στο μέλλον. Γιατί όλοι σας είστε υπεύθυνοι για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλοι σας είστε υπεύθυνοι για όλες τις αποφάσεις, θεωρητικά το λέω, των κρατών μελών και των κυβερνήσεών τους. Άρα ας μην ε, κάνουμε προσωπικές επιθέσεις αν θέλετε, μπορούμε να επικρίνουμε την πολιτική ορισμένων κυβερνήσεων. Μπορούμε να συζητάμε την πολιτική κυβερνήσεων, γιατί είμαστε κοινοβουλευτικοί. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, λοιπόν, να επικρίνουμε και να επιτιθέμεθα κατά κυβερνήσεων ή κατά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λυπάμαι, λυπάμαι που το λέω ακόμη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένε φορέ χρειάζεται, είναι απόλυτα αναγκαίο να την κατακρίνουμε και το ξέρετε. Αυτό κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα. Βλέπετε ότι όλη μας η συζήτηση μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν ιδιαίτερα πολιτική. σα. ευχαριστώ πολύ για την ε, συμμετοχή σας.